adopting the agenda. If there are no objections, you know the agenda, it is adopted with the following changes. Following a request by Yannick Jadot, item 9. Με τις ακολουθές αλλαγές, το σημείο 9 θα το αλλάξουμε με το σημείο 12 σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία. Θα πρότεινα να ψηφίσουμε πρώτα τα σημεία 4 και 5 και κατόπιν να τελειώσουμε με το σημείο 3. Θέλω να υποθυμίσω στα μέλη ότι οι αλλαγές στην ημερήσια διάταξη στο στάδιο αυτό μπορεί να έχουν συνέπειες ως προς την διαθεσιμότητα των εκπροσώπων της Κομισιόν ε, κατά τη συζήτηση των θεμάτων ε, και επίσης και των μελών προσκεκλημένων κλπ. Έτσι λοιπόν προσπαθήστε σας παρακαλώ στο μέλλον να κρατήσετε αυτές τις αλλαγές στο ελάχιστο. announcements, Λοιπόν, σημείο 2, ανακοινώσεις. Έχετε το κατάλογο στο φακελό σας, ε, ως συνήθως. Ε, υπάρχουν κάποιες αλλαγές βέβαια. Με, πολύ προσωπική ικανοποίηση θα παρουσιάσω την κυρία Ντοναντέλ Πίμπαλς, η οποία είναι, έχει διοριστεί ε, επικεφαλής ε, της Διεύθυνσης για τις σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ, Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού και από τον επόμενο Ιανουάριο θα αναλάβει τα καθήκοντά της. Ε, η Τεμετέλα έχει εργαστεί πάρα πολύ σκληρά από τη δημιουργία αυτής της Επιτροπής το 2004 και έχουμε όλοι εποφεληθεί από την εξαιρετική δουλειά της και από την αφοσίωσή της σε αυτή την Επιτροπή. Σίγουρα θα μας λείψετε εδώ στην Επιτροπή μας, Ντονατέλα. Σας ευχαριστώ συγχαρητήρια για αυτή την προαγωγή και ελπίζω ότι θα συμβάλλει η προαγωγή σας ε, για την ε, σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Σας προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Όπως σας είπα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το σημείο 4. σχετικά με την γνωμοδότηση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μαύρη Θάλασσα. Με την Κάζακ είναι ο εισηγητής. Τροπολογία 1, τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Πάλι τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ... Α, συγγνώμη, τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της 10. Πρώτο τμήμα της 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά αποχές Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 17 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 18. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή με συντριπτική πλειοψηφία. 20 υπέρ, μία ψήφος κατά. Συμπεριλήφθηκε η δική μου ψήφος. Συγχαρητήρια στον Μέτιν Κάζακ. Και πάμε στο σημείο 5. είναι η ψηφοφορία για την πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την χορήγηση ε, νοσιακή ε, εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ζημίε ε, από εγγυήσει και δάνεια για έργα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο William Dartmouth είναι ο εισηγητής και αρχίζουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 61 τμήματική ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ. Κατά κατά αποχές δεκτή. 32. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ έλεγχος Α, πάμε πίσω στην 64 για να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 Υπέρ του της 35 κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος στην 66 άρχεται η ψηφοφορία πέρας με την ψήφο μου ε, υπέρ απορρίπτεται όμως η τροπολογία 36 Δεν έχω την κάρτα, αλλά ψηφίζω υπέρ της 66. Ε, Οπότε είναι δεκτή. Η 66 λοιπόν έγινε δεκτή. Το ανακοίνωσα εγώ, ανακοίνωσα τη θετική μου ψήφο από πριν, πριν από το τέλος, τέλος της ψηφοφορίας. Παρακαλώ πολύ. Πάμε στην 36, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα πάμε στα εκτιμώντας. 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 2. Ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 τμηματική ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 τμήματική ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Α, έλεγχος. Ελέγχομαι το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγώ ψηφίζω υπέρ. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Υπέρα. Κατά αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 48. Υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. Τροπολογία 8. Ο κύριος Κάσπερη. Μια ερώτηση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της 48. Η 48, η 48 ε, ε, έγινε δεκτή ή όχι. Ναι, έγινε δεκτή. Ναι. Ψηφίστηκε 48. Πάμε τώρα στην τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41, όχι 51, 51 συγγνώμη, υπέρ της 51, κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία, την 51. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 9. Πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 14 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται, η 55 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται, 15 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 17 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Η 18 υπέρ, τη 17, άρχεται η ψηφοφορία για τη 17. Εγώ ψηφίζω κατά. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές Δεκτή. Έλεγχος. Ελέγχουμε την 56 τροπολογία. Εγώ ψηφίζω υπέρ, άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, εγώ ψηφίζω υπέρ. Και πέρας. Και εγκρίθηκε 21 ψήφισαν υπέρ Κανείς δεν ψήφισε κατά και έχουμε και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια στον William Dartmouth. Πάμε στο σημείο 3. Well, this is the this file, please. May I have your attention, please? Προσοχή, προσοχή, παρακαλώ είναι για το κοινοτικό σύστημα ελέγχου εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης. Ο εισηγητής μας είναι ο Γιώργ Λάιχτφριντ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Πρόσφατα θέλαμε να ψηφίσουμε το σχέδιο έκθεση σήμερα, είχε σχεδιαστεί, μετά από μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εισηγητού και σκιωδών. Παρακαλώ, τι πάθατε Έγιναν λοιπόν άτυπες συνομιλίες μεταξύ του εισηγητή και την Κομισιόν επίσης και ενημερώθηκα ότι θέλει ο εισηγητής να αναβληθεί σε άλλη συνεδρίαση ψηφοφορία. Αντί να ψηφίσουμε σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, ο εισηγητής θέλει να εξετάσουμε τις τροπολογίες ε, Όσοι ήθιστε στην Επιτροπή μας πρέπει να ζητήσω από τους συντονιστές αν συμφωνούν με την πρόταση αναβολής της ψηφοφορίας. Συντονιστές και Επιτροπή γενικότερα. Είστε υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας εδώ. Δεν ενίσταται κανείς. Εντάξει. Δίνω το λόγο λοιπόν στον Γιώργ Λάιχτφριντ ο οποίος θα κάνει μια εισαγωγή στις τροπολογίες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξηγήσω την πρόταση αναβολής ευθύς εξ αρχής. Ε, είχαμε ένα νομικό πρόβλημα ή τέλο πάντων δόθηκε εντύπωση ότι υφίστατο νομικό πρόβλημα, διότι εμείς και το Συμβούλιο Είχαμε ως αφετηρία διαφορετικούς τίτλους κανονισμών στις διαβουλεύσεις μας εμείς είχαμε την παλιότερη έκδοση, το Συμβούλιο είχε την νεότερη έκδοση και αυτό οδήγησε σε κάποια βεβαιότητα αν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Κάναμε μακρές διαβουλεύσεις, αλλά συνεχίζαμε και τις εργασίες μας. Δηλαδή, ετοιμάσαμε σχέδιο έκθεσης, υπάρχουν και τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για το σχέδιο έκθεσης αυτό. Παράλληλα όμως με την Κομισιόν είχαμε εντατικέ επαφές για να δούμε πώς θα εξομαλύναμε τα πράγματα. Μετά προέκυψε η δυνατότητα να προχωρήσουμε βράχη πρόθεσμα να πρόθεσμα δηλαδή να απορριφθεί η πρόταση της Κομισιόν από την Επιτροπή και θα υπήρχε η δυνατότητα η Κομισιόν να αντιδράσει γρήγορα ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις στην κατάθεση νέας πρότασης στο Κοινοβούλιο. Αυτή η δυνατότητα για κάποιο διάστημα θεωρήθηκε πολύ εφικτή, αλλά στο τέλος διαπιστώσαμε ότι αυτή η διαδικασία, όπως την είχαμε υπόψη μας, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Παράλληλα εσείς κύριε Πρόεδρε και η Επιτροπή έτσι απευθύ... Ε, λάβατε επιστολή από τον αρμόδιο Επίτροπο όπου η Κομισιόν διαπιστώνει ουσιαστικά ότι η διαδικασία μας ως έχει είναι σωστή. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει για μας το εξής ότι εγώ μαζί με τους ε, σκιώδεις αποφασίσαμε να δώσουμε συνέχεια στις εργασίες μας και γι' αυτό όμως χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος από τον προβλεφθέντα. Όλη η θεματική δεν είναι τόσο περίπλοκη στις επιπτώσεις της, αλλά με όλα αυτά τα μπερδέματα και με όλες αυτές τις διευρύνσεις των δυνατοτήτων που έχουμε στα πλαίσια της γενικότερης λύσης που εξέβραμε, δεν ήταν τέλος πάντων μετά από όλα αυτά δυνατόν να προλάβουμε να συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες, να πούμε ποιο το καλό, ποιο το κακό και νομίζω ότι αν θέλει κανείς να καταλήξει σε ένα καλό αποτέλεσμα απαιτείται περισσότερος χρόνος. Αυτό ήταν απαραίτητο. Με την αναβολή του όλου θέματος δεν δημιουργείται και μεγάλο πρόβλημα γιατί το σύστημα κατά το ίμιση λειτουργεί ούτως ή άλλως τώρα. Και με όλους τους εμπλεκομένους κάναμε συζητήσεις και δεν υπήρξαν μεγάλες επιφυλάξεις σε σχέση με την αναβολή της ψηφοφορίας αν προκύψει ένα αποτέλεσμα καλό μετά από όλα αυτά. Και περνάω στην ουσία. Τι λοιπόν ε, είναι, τι θα είναι ε, ε, πότε θα είναι καλό να βρούμε ένα σύστημα το οποίο θα δημιουργήσει ενία πρότυπα στην Ευρώπη για την εξαγωγή αυτών των διπλής χρήσης ειδών, να μην υπάρχουν τόσες διαφορές όπως τώρα, να είναι διαφανές το σύστημα, να είναι ένα σύστημα όπου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να παρεμβαίνει στον έλεγχο με μορφή που θα συζητήσουμε ποια θα είναι και νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε κάποια αντικείμενα, κάποια θέματα τα οποία δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο σύστημα μετά από νεότερες εξελίξεις στον τομέα της σύγχρονης μορφής, αν θέλετε, αντιπαράθεσης θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. Πρόσφατα ακούσαμε ότι κάποια κράτη ισχυρίστηκαν ότι αντιμετωπίζουν επιθέσεις. Ε, μπορεί να υπάρξει σαμποτάζ πυρηνικών εργοστασίων, για παράδειγμα. Ε, αυτό είναι κάτι πολύ δυσάρεστο, αν δεν μπορούν να αντιδράσουν οι άνθρωποι εκεί επί τόπου. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε και για όλα αυτά απαιτείται περισσότερος χρόνος. Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους κυρίους Κασπάρη και Στέρντι ως επιτοπλίστων είναι, θεωρώ, τροπολογίες που σε μεγάλο βαθμό ε, μπορούν να ενταχθούν στο γενικότερο πλαίσιο. Υποθέτω, θα τα ξέρουμε αυτά στο τέλος της συζήτησης, ε, θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε μια λογική πρόταση, αλλά για να δουλέψουμε με ακρίβεια και όσο γίνεται καλύτερα, θα παρακαλούσα την Επιτροπή και εσάς κύριε Πρόεδρε θα σας παρακαλούσα λοιπόν να γίνει τον Ιανουάριο η ψηφοφορία, γιατί δεν προλαβαίνουμε τον Δεκέμβριο. Ε, καλύτερα να δώσουμε λίγο χρόνο, ούτως ώστε να είναι στέρεο το αποτέλεσμα και καλό. Ευχαριστώ. Όπως ε, γνωρίζετε, έχουμε λάβει την επιστολή από τον Επιτροκό Ντικούχτ και αντιμετωπίζεται εκεί στο νομικό πρόβλημα που έθεσε ο εισηγητής και λέει ότι δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της πρότασης. Έτσι λοιπόν, πριν να ανοίξω τη συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, ίσως θα πρέπει να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Παύλο για το θέμα αυτό, αλλά και επί της ουσίας των ε, τροπολογιών που προτείνονται από τον κύριο Συγητή. Παρακαλώ, πού είστε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι ευχαριστώ τον συγητή για το εξαιρετικό, του, το εξαιρετικό του έργο για το θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα θέμα όπου υπήρχε ένα θεσμικό νομικό πρόβλημα και δεν το είδαμε από την αρχή ε, όταν ε, διαβιβάστηκε η στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει κανονισμού του 2000 κατόπιν τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο το 2009. Το καλό με το πρόβλημα αυτό είναι ότι το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με την υιοθέτηση και τη θέση σε σχήμα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι λοιπόν ε, δεν είναι κάτι που θα ανακύπτει συχνά στο μέλλον. Είναι άπαξ πρόβλημα. Έτσι λοιπόν χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι έχει την καλοσύνη ο εισηγητής να υιοθετήσει την πρόταση που έγινε από τον Επιτροπό μας. Δηλαδή, να μπορέσει η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να τροποποιήσουν τον ε, τίτλο του κανονισμού και να προχωρήσουμε με τις τροπολογίες. Ε, χρειάζεται περισσότερος ε, χρόνος, συμφωνούμε, είναι πολύ πλοκό το θέμα για τις τροπολογίες Έχουμε ε, το θέμα των προϊόντων και έχουμε κάποια τροποποίηση σε σχέση με τις χώρες. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες για την εισαγωγή και την καταχώρηση και αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε αν ε, χρειάζεται συμβουλή της Κομισιόν από αυτό ο στόχος της Κομισιόν είναι ίδιος με το στόχο του εισηγητή, δηλαδή να έχουμε ένα καθεστώς διαφανές μίσους κανόνες για όλους τους εξαγωγείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όσο το δυνατόν λιγότερο διοικητικό άχθος για τους εξαγωγείς μας, ε, έτσι ώστε αφενός ε, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που ενίοτε έχουμε με αυτά τα προϊόντα. Ξέρουμε ότι είναι τα πιο αναπτυγμένα τεχνολογικά προϊόντα και επί αφετέρου το θέμα της ασφάλειας που αποτελεί τη βάση όλων αυτών. Κάποιο είπε ότι ο καλύτερο τρόπο να κάνουμε τον ελέγχο ε, είναι να έχουμε έναν υψηλό φράχτη. Ε, έτσι λοιπόν εδώ προσπαθούμε να ε, διατηρήσουμε τις λιγότερο δύσκολες και ευαίσθητες συναλλαγές ε, σε αυτό το κοινό σύστημα άδεια γενικευμένων εξαγωγών. Έτσι λοιπόν ε, θεωρούμε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να επιληθεί αυτή η νομική παρεξήγηση και υποστηρίζουμε λοιπόν τη λύση που προτάθηκε από τον συγητή. Αν υπομονούμε να συζητήσουμε επί της ουσίας τους επόμενους δύο μήνες. Ε, συμφωνούμε ότι ο Ινάριος είναι μια καλή χρονική στιγμή για την ψηφοφορία. Δύο μήνες καθυστέρησης δεν θα παρουσιάσει μεγάλο πρόβλημα. Κινείται βέβαια ο φάκελος, ε, σημειώνεται πρόοδος και σε αυτή την επιτροπή έχει δηληφθεί η πρόταση τροποποίηση του παραρτήματο 1 του ίδιου κανονισμού με αυτό που σχετίζεται με το κατάλογο των προϊόντων που θα ελέγχονται και η ανακοίνωση της Κομισιόν ε, για ε, το εμπόριο έχει δημοσιευθεί ήδη σήμερα και θα δείτε ότι υπάρχει και μία συνιστόσα για τους εξαγωγικούς ελέγχους ε, για τα προϊόντα διπλής χρήσης. Έτσι λοιπόν είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και στο μέλλον και ανυπομονούμε φυσικά να έχουμε το ίδιο καλό πνεύμα συνεργασίας που είχαμε μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Okay. Uh, thank you for your... Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Θέλει κανείς το λόγο. Κύριε Κάσπαρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, δύο παρατηρήσεις έχω. Καταρχήν για το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει μεγάλη κατανόηση και ασχολείται με το θέμα αντί να απορρίψει και η επιστολή του Επιτρόπου στην ε, Επιτροπή υπό όρους βοηθάει. Δεν είναι απόλυτα αιτιολογημένη. Οι επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα και εμείς έξι μήνες τώρα ασχολούμεθα με το θέμα είπαμε ότι έχουμε δυσκολίες, το είπαμε από την αρχή ότι είναι παλιά η νομική βάση, είναι πεπαλαιωμένος ο φάκελος που μας δόθηκε και η Κομισιόν είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή της. Έξι μήνες συγκεκριμένα για να επεξεργαστεί την πρόταση και να μας δώσει ενημερωμένη πρόταση και νομίζω ότι η Κομισιόν δεν έκανε σωστά τη δουλειά της Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι δείχνει μεγάλη κατανόηση το Κοινοβούλιο και όχι προς την Κομισιόν, αλλά προς τις επιχειρήσεις που πρέπει να έχουν ένα νομικό πλαίσιο. Εμείς μιλάμε εδώ για πολύ ευαίσθητα προϊόντα. Παρακαλώ τους συναδέλφους όμως να λάβουν υπόψη ότι δεν μιλάμε για ε, τεθωρακισμένα ή πυράβλους, που θα μπορούσαν να έχουν και πολιτική χρήση και γι' αυτό είναι, τα λέμε διπλής χρήσης. Μιλάμε για στάνταρ κλασικά προϊόντα, φορτηγά, υπολογιστές και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται ως επιτοπλίστων ε, για ειρηνικούς σκοπούς. Την κατάχρηση θα πρέπει να εμποδίσουμε και γι' αυτό παρακαλώ να το εξετάσουμε το θέμα με την ησυχία μας και γι' αυτό συμφωνώ με τον εισηγητή και υποθέτω ότι μέχρι τον Ιανουάριο θα έχουμε μια ευρεία πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης εδώ στην Επιτροπή. Αλλά ξεκολουθείτε να πιστεύετε ότι ε, το, η σωστή θέση είναι να αναδιατυπώσουμε την πρόταση. Όχι. Μάλιστα. Ο κύριος συγητής θέλει να επανέλθει. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλα υπόθηκαν για σήμερα. Και τώρα πρέπει να αρχίσουμε τη δουλειά και να σταματήσουμε τα λόγια. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ας περάσουμε στο σημείο 6, σύμφωνα με τις αλλαγές που κάναμε. Στην ημερησία διάταξη, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Κορέας. Εδώ θα εξετάσουμε σχεδίο έκθεση που έχετε στο φακελό σα. Εισηγητή είναι ο κύριο Ρομπερτ Στάρτη από το ECR. Εδώ υπάρχει αντίθεση σε σχέση με το όσα διαβάσαμε στα μέσα μαζική ενημέρωση τι τελευταίε εβδομάδε, ε, Δεν φταίει το Κοινοβούλιο που κύρωσε αυτή τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών έχει καθυστερήσει. Αντίθετα, όπω ξέρετε, έχουμε ξεκινήσει τι διαδικασίε και ξεκινήσαμε να εξετάζουμε τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών πολύ νωρί, ε, χωρί καν να έχουμε λάβει την επίσημη παραπομπή από το Συμβούλιο. Και γι' αυτό εγώ αισθάνθηκα ότι θα έπρεπε να διορθώσω αυτές τις λεθασμένες πληροφορίες ε, που δημοσιεύτηκαν από τους Financial Times και έτσι διένυμα την επιστολή μου, η οποία δημοσιεύτηκε από τους Financial Times. Έτσι λοιπόν, να δώσω τώρα το λόγο στον συγητή, τον κύριο Στάρντι. Πού είστε? Uh, Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να σχολιάσω την επιστολή σας και θέλω να σας ευχαριστήσω τα γιατί εμείς ήμασταν ε, σε συζητήσεις και τώρα η κατάσταση ε, οδεύει προς ολοκλήρωση. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω ε, πολλούς. Όμως έστειλα και την δήλωσή μου σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου και ελπίζω να είχαν την ευκαιρία να τη διαβάσουν και να τη χωνέψουν. Τον Απρίλιο του 2007 τα κράτη-μέλη επέτρεψαν στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί μια φιλόδοξη και πλήρη συμφωνία ελευθερών συναλλαγών με την Νότιο Κορέα. Μετά από οκτώ γύρου επίσημων διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές μονογράφησαν τη συμφωνία τον Οκτώβριο του 2009 και έτσι όσο μόλι είπατε αρχίσαμε να εργαζόμαστε πολύ νωρίτερα για το θέμα αυτό. Είσαι, αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικό εμπόριο σε γεωργικά, βιομηχανικά αγαθά και στι υπηρεσίες παρά τα προφανή αναμενόμενα ωφέλη η συμφωνία θα φέρει ε, που θα φέρει στους καταναλωτές. Ε, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ε, η συμφωνία έχει μόνο ονομαστική αξία. Η Ευρωπαϊκή πρέπει να δοθεί μάλλον μια έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών βάσει της συνθήκης Λισαβόνας και πρέπει να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι το καθήκον μας να κάνουμε συστάσεις για το κείμενο αλλά να έχουμε μια προσέγγιση ωφέλους και ε, να δούμε αν είναι στο σύνολο, προς όφελος της κοινότητας στο σύνολό τη ε, να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποιες τροπολογίες, απλώς μια σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της συμφωνίας. Ε, Παρ' έχουμε μια ρήτρα διασφάλισης και θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και του άλλου και συζητητέ που εργάστηκαν σκληρά για την έκθεση αυτή. Η δέσμευσή του στη διαδικασία του τριμερούς διαδιαλόγου ε, και ε, η δική σας ηγεσία, Πρόεδρε, μα βοήθησε στο να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και διατηρούμε τη δέσμευσή μας ε, για να ενισχύσουμε τι σχέσει με τους Νότιους Κορεάτες. Η ρήτρα αυτή έχει να κάνει με πάρα πολλά θέματα όπως έχουν να κάνουν η εποπτεία, η παρακολούθηση, η υποβολή αναφορών, επιτροπολογία, ο ρόλος των θεσμών, ε, η επιστροφή δασμών κτλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον Πρόεδρο για τη θέση του για την, στην επιτροπολογία. Ε, ότι έχετε νομικές γνώσεις ως δικηγόρος. Ε, ήταν ε, κάτι πολύτιμο για αυτή την Επιτροπή και πάλι σας ευχαριστώ. Εγώ έχω εκφράσει στο επεξηγηματικό κείμενο τη θέση μου με πολλές λεπτομέρειες και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τις συστάσεις που έχετε στείλει για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής σε ένα ζήτημα ε, για τις προτάσεις ε, για το διοξείδιο του άνθρακα της Νοτιού Κορέας το σχέδιο νομοθεσίας αν εγκριθεί ως έχει θα μπορούσε να επιβάλλει δυσανάλογο άχθος στους Ευρωπαίους ε, ε, εξαγωγής αυτοκινήτων ε, οι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα των αυτοκινήτων που εξάγουν στη Νότια Κορέα αλλά δεν μπορούμε να τους ζητάμε εδώ να κάνουν μεγαλύτερη μεγαλύτερες προσπάθειες ε, από τους νοτιοκροατές, γιατί κάτι τέτοιο θα έχει αρνητική ε, επίπτωση στον ανταγωνισμό. Ε, προετοιμάζεται μια διαβούλευση με την βιομηχανία, με τον τομέα για να δούμε τα πιο σημαντικά στοιχεία των εκπομπών για το διοξίδιο του άνθρακα και της νομοθεσία Θέλουμε να έχουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν και την προστασία του περιβάλλοντος επίση θέτουμε θέματα που αφορούν ε, το σχέδιο νομοθεσία ε, για το πλαίσιο, ε, για την ποιτή, για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Ε, μέχρι το τέλος ε, του έτους ε, πρέπει να έχει υιοθετηθεί νομοθεσία η Κομισιόν παρακολουθεί αυτό το θέμα έτσι ώστε να μην τεθούν τεχνικά εμπόδια για το εμπόριο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των αυτοκινήτων των Ευρωπαίων εξαγωγέων στην αγορά της Νοτιού Κορέας. Μπορεί να έχει αλλάξει η κατάσταση τώρα, αλλά πρέπει να το θέσουμε αυτό το θέμα και να το βάλουμε στην έκθεση γιατί ε, έπρεπε να μεταφραστεί και έτσι λοιπόν ε, έχουμε εδώ τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά και εδώ ε, θέλουμε να εμπλακεί ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανία στο διάλογο της Κομισιόν με τους Νότιο Κορεάτες. Αναγνωρίζουμε εδώ ότι σε ορισμένους ε, τομείς ε, αν οι Κορεάτες μετακινηθούν προς τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τότε θα έχουμε αμοιβαία ωφέλη. πρέπει να έχουμε ένα συνεχή διάλογο και όχι κάτι που θα αφαιθεί στα γραμματοκιμώτια των μελών αυτής της Επιτροπής. Εγώ συνεργάστηκα πάρα πολύ πολύ σκληρά και πολύ στενά με τους συναδέλφους στην Κομισιόν για να θέσουμε τα θέματα επιτάπητος πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Καλούμε την Επιτροπή να δώσει επαρκή χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει επαρκώ την πρόταση και οποιοδήποτε αντίκτυπο μπορεί να έχει στην ε, συμφωνία. Ε, η τακτική διαδικασία έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2011. Πρόεδρε, όπω είπα και στην αρχή, όλοι έχουν αντίγραφο ε, της ε, δήλωσής μου και θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλια αυτή τη Επιτροπής. Σα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ. Νομίζω ότι αιτιολογείται πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα μέλη ε, της Επιτροπής, να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προβλήματα που έχουν τεθεί από τον εισηγητή. Κύριε Γκαρσία, παρακαλώ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Πριν αναφερθώ στα θέματα που αναφέραν από τον κύριο Στάρτη, να πω από την πλευρά της Κομισιόν πόσο εκτιμούμε την εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για το φάκελο της Κορέας και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και σε ό,τι αφορά τη σύνοψη τη σχέση. Νομίζω από την αρχή τη διαδικασία ο Επιτρόπο Δεγκούχτε είπε με σαφήνεια ότι ε, η συμφωνία θα ε, υπογραφεί και θα εφαρμοστεί κατόπιν τη ε, εξέταση και έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτή ήταν η σωστή στάση που έπρεπε να ακολουθηθεί και νομίζω ότι με πολύ υπευθυνό τρόπο διαχειρίστηκε το φάκελο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό το καλωσορίζουμε σε ό,τι αφορά τώρα τον κανονισμό για το δεξίδι του άνθρακα. Θα ήθελα να διασφαλίσω όλα τα μέλη της Επιτροπής ότι παρακολουθούμε αυτό το θέμα πολύ στενά ξεκαθαρίσαμε στις κορεάτικες αρχές ότι ορισμένες ε, πτυχές του σχεδίου θέτουν ε, δυσανάλογο βάρος στους Ευρωπαίους εξαγωγείς και επίσης διαβουλευόμαστε πολύ στενά και με τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Όταν θα ολοκληρώσουμε το έγγραφο που προετοιμάζουμε θα το στείλουμε στις κορεατικές αρχές για να τους πούμε ποιες πτυχές αυτού του κανονισμού πρέπει να αλλάχθουν κατά τη δική μας άποψη και ευχαρίστω να γνωστοποιήσω αυτό το εγγραφό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και βέβαια υπάρχουν κάποιες απαιτήσει εμπιστευτικότητα, αλλά μπορώ να σα διαβεβαιώσω το εξή, ότι τη στιγμή που ε, ο κανονισμός ε, θα δημοσιευθεί από τους Κορεάτες, στην οριστική του μορφή, θα κάνουμε μια προσεκτική εξέταση και θα σας γνωστοποιήσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα κράτη-μέλη πριν να προχωρήσουμε περαιτέρω στο θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, ευχαρίστως ε, μαζί με την Επιτροπή να κάνουμε μια αξιολόγηση του κανονισμού. Και θα ξεκαθαρίσουμε στους Κορεάτες ε, συναδέλφους ότι ορισμένες πτυχές αυτού του κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθούν για να μην επιβληθεί αυτό το άχθος ε, ε, στους Ευρωπαίους εξαγωγείς. Θα περιοριστώ εδώ, αλλά αν υπάρχουν ερωτήσεις από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευχαριστώ να απαντήσω. Thank you. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω πιστεί ότι πρέπει να πούμε χωρίς άλλο ναι στην ε, συμφωνία, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά. Ένα πρόβλημα το είπατε κι εσείς, εγώ έχω κι άλλα. Με τη συμφωνία αυτή θα έχουμε ένα ε, νομοθέτημα που δεν θέτει επίσης όρις όλους τους ε, κλάδους της βιομηχανίας. Παίρνουμε την αυτοκινητοβιομηχανία. Υπάρχει δυνατότητα η κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία να αξιοποιεί από τρίτες χώρες ε, εξαρτήματα. Αυτό είναι ένα θέμητο πλεονέκτημα υπέρ της βιομηχανίας τους. Όταν πρόκειται δηλαδή για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπορεί ο Κορεάτης ε, να πάρει αδασμολόγητες μπαταρίες, μπαταρίες από, την Κίνα, από και να τις ενσωματώσει, ενώ ο Ευρωπαίος θα πρέπει να πληρώνει δασμούς. Οπότε αυτό μας δημιουργεί προβλήματα και στενοχώρια. Αυτά βέβαια έχουν ληφθεί εν μέρη υπόψη σε ό,τι αφορά το, την ε, ε αυτορύθμιση και εδώ έγινε μία ε, προσπάθεια εξέβρεση συμφωνίας και ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε που ακολουθήσατε ε, πολύ αυστηρά την επιτροπολογία. Αν όμως δω γενικότερα το θέμα και λάβω υπόψη μου και κάποια ε, θέματα που έχουν συμφωνηθεί αλλά δεν εφαρμόζονται, αναρωτιέμαι αν μπορούμε ανεπιφύλακτα να πούμε ναι. Ένα πρόβλημα είναι πράγματι τα μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο. Ο κύριος Στέρντι εδώ παρουσίασε την προβληματική. Αν τα δούμε όλα αυτά, διαπιστώνουμε σαφέστατα ότι η νομοθεσία για το διοξίδιο του άνθρακα είναι προς το συμφέρον των κορεατών βιομηχανιών. Πότε θα πάρει κανείς πιστώσεις, για παράδειγμα ούτως ώστε να επιτύχει κάποιες, κάποιους ευνοϊκούς όρους. Εκεί αποκλείονται οι Ευρωπαίοι ή οι διάφορες ε, ε κατατάξεις ε, του ε, βάρους. Αυτά είναι σε βάρος των Ευρωπαίων αυτοκινητών βιομηχανιών. Οπότε ενδεχομένως ε, θα αμφισβητηθεί μέσα από την η κειμένη νομοθεσία η συμφωνία. Υπάρχουν και άλλοι τομείς προβληματικοί. Ένας που με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι το θέμα των κοινωνικών προτύπων. Στο κεφάλαιο 13 έχουμε συμφωνήσει ότι θα, έχουμε, ε, θα δεχτούμε και θα εφαρμόζουμε τους βασικούς κανόνες του, ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας τρέχουν οι διαπραγματεύσεις με τους Κορεάτες ήδη, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει επιτελεστεί πρόοδο στη Νότιο Κορέα σε ό,τι αφορά δύο βασικά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Είναι η ελευθερία του συνεταιρίζεστε, που έχει συμφωνηθεί από το 1948 και είναι το πρότυπο 87, και η άλλη για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η 98, η οποία συμφωνήθηκε το 1949 και τα δύο πρότυπα η Νότια Κορέα δεν τα έχει επικυρώσει. Οπότε και ιδιαίτερα αν δούμε και την ανταγωνιστικότητα των Γερμανών, των Ευρωπαϊκών τέλος πάντων, των Γαλλικών βιομηχανιών, εδώ έχουμε κάποια βασικά θέματα που διαταράσσονται ε, άμα συγκρίνουμε τις, τους δύο τρόπους παραγωγής. Μέσα από κοινωνικό διάλογο δημιουργούνται άλλες συνθήκες ανταγωνιστικότητας από ότι αν δεν υπάρχει ο διάλογος ή και τα πρότυπα. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει κάποιος ευσεβής πόθος που περιλαμβάνεται στην συμφωνία και που δεν εφαρμόζεται όμως στην πράξη. Άρα θα ήθελα κάποιες σαφές, θα απαιτούσα σαφείς δηλώσεις από την κορεατική πλευρά, ώστε οι προθέσεις που έχουν υπογραφεί στη συνθήκη να έχουν και πραγματική ισχύ και να εφαρμόζονται στην κορεατική από την κορεατική νομοθεσία. Και τότε μπορούμε, χωρίς να μας τύπτει η συνείδηση, να ε, προσυπογράψουμε τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο κ. Ευχαριστώ. Εγώ μιλάω εξ ονόματος ε, του συναδελφού Τσαλένσκι, γιατί είναι καθοδόν. Καταρχήν ε, θα ήθελα να αυτή τη συζήτηση να την έχουμε κάνει αφού θα είχε εγκριθεί η ρήτρα και έχοντας όλα τα στοιχεία στη θέση μας στη στιγμή της αξιολόγησης αιτιολογικής έκθεσης του κυρίου Στάρμπη. Όπως είπε ο κύριος Στάρμπη, Υπάρχει μια σειρά θεμάτων ε, που είναι ανοιχτά ακόμη. Επιτροπολογία, ελπίζουμε να επιληθούν το συντομότερο δυνατόν και είμαστε φυσικά αισιάδοξοι το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν θα ξεκινήσει μια έρευνα το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα με τους Κορεάτες. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Παρ' όλα αυτά ευχαριστώ τον κύριο Στάρντι για το έργο του και τους σκιώδεις εισηγητές και εγώ νομίζω ότι είναι επιτυχής η εργασία όλων ε, των μελών της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου σε ό,τι αφορά τη ρήτρια διασφάλισης. Ελπίζω ότι αυτή η καλή δουλειά που υλοποιούμε και που ακόμη ε, πρέπει να επιτελέσουμε να είναι καρποφόρος και Φυσικά όλοι θέλουμε να πετύχουμε μια καλή συμφωνία. Πάντως επιμένω ότι ακόμη υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά ζητήματα, όπως είπε και ο συνάδελφο, ε, που πρέπει να ξεκαθαριστούν πριν να λάβουμε οριστική θέση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφος Βέρνερ Λάγκεν, γιατί θεωρώ ότι στην έκθεση του εισηγητή πολύ σωστά τίθενται ορισμένα θέματα, καθίσταται όμως σαφές ότι αυτά που βρίσκονται επί τάπητος δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές προκλήσεις. Στην τελευταία ε, συζήτηση, στην ευρίαση της Επιτροπής δεχτήκαμε τρεις σημαντικές εκθέσεις για το την προστασία του κλίματος και τις κοινωνικές ευθύνες και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και αναφέρονται δύο σημαντικοί για μένα τομείς, σημαντικοί και για την ομάδα μου, σχετικά με την προβληματική του σε ποιο βαθμό οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών απαντούν, συνιστούν μια γέφυρα για να απαντηθούν σοβαρά θέματα. Δηλαδή, το εμπόριο και η ανταλλαγή συγκεκριμένων αγαθών μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης, βελτίωση των κοινωνικών δικαιωμάτων για τους απασχολουμένους σε όλους τους τομείς της ε, εθνικής, των εθνικών οικονομιών και πώς μπορεί να συμβάλλει και πλέον στην προστασία του κλίματος. Οπότε θα πρέπει εδώ, σε αυτό το σημείο καμπή που φάσαμε, σε αυτό το σταυροδρόμι, να απαντήσουμε και αυτά τα θέματα και να ανταποκριθούμε και σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Από ό,τι γνωρίζω και από την συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά και από την προσέγγιση του εισηγητή, νομίζω ότι εδώ υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο τομείς. Ξέρουμε ότι η δημοκρατία της Νότιας, η Νότια Κορέα, Μόλις το Δεκέμβριο ψήφισε στο Κοινοβούλιο, όχι θα ψήφισε το Δεκέμβριο την νομοθεσία για το διοξίδιο του άνθρακα, άρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει το Κορεατικό Κοινοβούλιο πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν είναι σοβαρό το ζήτημα και πράγματι θα πρέπει να το ξαναδούμε. Μπορούμε ήδη με την ε, διατύπωσή μας ε, να προχωρήσουμε με τρόπο οριστικό, χωρίς να ξέρουμε τι θα κάνει τελικά η κορεατική πλευρά. Δεύτερον, τα βασικά πρότυπα εργασίας του ILO, του, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που ακόμα δεν έχουν κυρωθεί από την Κορέα. Ε, θα πρέπει πρώτα να κυρωθούν πριν αποφανθούμε υπέρ αυτής της συμφωνίας διότι δυστυχώς ξέρουμε από το παρελθόν ότι συχνότατα οι δηλώσεις προθέσεων παραμένουν δηλώσεις και δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ρωτήσουμε την Κομισιόν σε ποιο βαθμό στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την κορεατική πλευρά θα επιμείνουν στην υποχρέωση τήρησης των προτύπων, ώστε να καταστεί σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ θα περάσει σε μια νέα κατηγορία συμφωνιών με τις βιομηχανικές χώρες, ε, τις τρίτες χώρες ε, και θέτει θέματα κοινωνικά, θέματα προστασίας του κλίματος και θέματα απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει τώρα να προχωρήσουμε. Ο κύριος Κάσπαρη από το ΕΛΚΑ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ε, νομίζω ότι μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων μπορούμε συγκεκριμένα να φροντίσουμε την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Καλό πράγμα αυτό. Ε, πριν από χρόνια θεωρούσαμε ότι θα ήταν καλό με αυτόν τον σημαντικό εταίρο να συνάψουμε μια τέτοια συμφωνία. Ξέρω με τα θέματα του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα είναι μια δοκιμή, μια λιδία λίθος με τους Κορεάτες, αν δηλαδή θα προχωρήσουν οι Κορεάτες. Ε, ελπίζω ότι η νοτιοκορεατική πλευρά με τρόπο συνειδητό θα προχωρήσει. Αλλά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, εμείς τα τελευταία χρόνια περάσαμε την νομοθεσία για το διοξίδιο του άνθρακα και στα, στα φορτηγά και τώρα πάμε στα αγιοταχή. Ξέρουμε ότι δεν γίνεται δεκτή κάθε πρόταση από την Κομισιόν, ε, τροποποιείται από το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι η... Ε, στην βιομηχανια υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Θα ήταν πολύ άσχημο. να ε, απαιτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αλλάξει άρδιν την τροπολογία ε, προς όφελος της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ε, υπάρχουν και σε σχέση με τους Κορεάτες κάποιες βελτιώσεις, χρειάζονται, θα πρέπει να γίνουν, καλό είναι και σημαντικό είναι να αυξήσει και τις πιέσεις η Κομισιόν προς τους Κορεάτες, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ξέρουμε ότι το υπέρ ή κατά σε μια τέτοια συμφωνία δεν θα εξαρτηθεί από το αν θα χαρεί η αυτοκινητοβιομηχανία σε τελευταία ανάλυση, διότι ανεξάρτητα από το τι μορφή θα έχει η νομοθεσία για το διοξείδιο του άνθρακα στην Κορέα, ποτέ η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα είναι ευχαριστημένη απόλυτα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον ω κοινοβούλιο το θέμα, ώστε να βρούμε τη σωστή ισορροπία και τη σωστή λύση στο θέμα. Τώρα, για τα πρότυπα εργασία, τα βασικά πρότυπα τη ΔΟΕ. Είναι σημαντικό να τηρηθούν κάποια ελάχιστα πρότυπα. Πιστεύω ότι έχουμε συμφωνήσει ότι μια διαπραγματευτική συμφωνία σημαίνει ότι δεν θα αρχίσουν από την πρώτη μέρα να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Οπότε συμφωνώ ότι εδώ θα πρέπει να συνεχίσουμε τις πιέσεις σε αυτό το τομέα, αλλά να ξέρουμε από την άλλη πλευρά ότι και εμεί από η ευρωπαϊκή πλευρά ε, ορισμένες προθεσμίες δεν τις ε, τηρήσαμε από την πρώτη μέρα που τέθηκαν σε ισχύ. Ε, έχουμε προβλέψει πολλές φορές μεταβατικές περιόδους πενταετούς διάρκειας ώστε η βιομηχανία, η, τα διάφορα συμφέροντα να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Οπότε είναι αυτονόητο ε, να προβλέψουμε και για τους Κορεάτες ένα τέτοιο διάστημα, μια τέτοια προθεσμία. Στις διαπραγματεύσεις με τους Κορεάτες, ίσως για πρώτη φορά υπάρχει κοινή επιτροπή μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαμε να έχουμε μια επιτροπή μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κορεατικού Κοινοβουλίου, όπως είχε ζητηθεί και για άλλε ε, ε, εκθέσεις, ούτω ώστε να υπάρχει κοινή επιτροπή, εκτός από την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου και την αρμόδια επιτροπή στο Νότιο Κορεατικό Κοινοβούλιο, ώστε οι επιτροπές ε, ε, να μπορούν να ε, συνεδριάζουν από κοινού μια φορά το χρόνο τουλάχιστον και να διαπιστώνεται από τα κοινοβούλια ότι τηρούνται οι συμφωνίες και αν δεν τηρούνται θα πρέπει να καλείται η Κομισιόν να προβαίνει στα απαραίτητα μέτρα. Σε ό,τι αφορά τα ανοιχτά θέματα, τα μη εμπόδια στο εμπόριο, ε, υπάρχει νομοθεσία ε, η οποία θα εγκριθεί από την Κορέα αλλά και από εμάς, διότι και εμείς μπορούμε να λάβουμε μέτρα, ώστε να δώσουμε συνέχεια να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Τέλος, δεν είμαι ευχαριστημένο, καθόλου ευχαριστημένο ε, από μια απόφαση του Συμβουλίου που λέει ότι η προσωρινή εφαρμογή ε, τη συμφωνία στην 1η Ιουλίου θα εξαρτηθεί από το αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα, θα έχει δώσει την έγκρισή του στη συμφωνία. Δεν λέει στην απόφαση ότι εμείς είμαστε υπέρ μιας προσωρινής εφαρμογής, αλλά λέει ότι το Συμβούλιο την 1η Ιουλίου θα αφήσει να τεθεί σε ισχύ η προσωρινή λειτουργία, εάν, την προσωρινή εφαρμογή, συγγνώμη, εάν έχει αποφανθεί θετικά υπέρ της συμφωνίας στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά του μηχανισμού διασφάλιση, Θα πρέπει να βρούμε μέχρι 30 Ιουνίου μια λύση. Ίσως και η νομοθεσία ε, για το διοξείδιο του άνθρακα να έχει ολοκληρωθεί στην Κορέα. Το προβλέπει το χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ ε, θετικό από το Συμβούλιο να θέτει υποπίεση το Κοινοβούλιο. εμεί έχουμε άλλη συμφωνία και σε μια ακρόαση εδώ στην Επιτροπή και νομίζω ότι ο Επίτροπος θα πρέπει να σκεφτεί μήπως θα πρέπει να καταστήσει σαφές στο Συμβούλιο ότι δεν είναι καθόλου φιλικό προς την Κομισιόν και την, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν θέτει, όχι, όχι ένα αμφιβόλ, όχι, ίσως να θέτει ένα αμφιβόλο για να μην μπορεί να υπονομεύει τις συμφωνίες που έχουν συναυθεί με το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να επιλέξει ο Επίτροπος μια διαφορετική προσέγγιση. Ε, είναι και θέμα ύφους, αν θέλετε, ε, στις συναλλαγές μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ή Συμβουλίου και Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορώ να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γκάσπαρη είναι εισηγητής εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για μια γνωμοδότηση. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ένα από τα πιο σημαντικά ε, μέσα στις, ε, ε, στους στόχους της Επιτροπής στην αρχή των προσπαθειών της αυτή τη φάση. Για το ελεύθερο εμπόριο πρέπει να πούμε ότι πάντοτε είναι ωφέλιμο προς τον καταναλωτή και ότι παρέχει πάντοτε ε, σταθερές αξίες. Ε, πρέπει να πούμε ότι 7 από τους διακεκριμένους ε, συναδέλφους μου θεώρησαν ότι αυτή η συνθήκη για το εξωτερικό εμπόριο αποτελεί, δίνει πολλούς φραγμούς και θέλησαν να κάνουν αλλαγές και να θέσουν ορισμένα εμπόδια στην εμπορική συμφωνία. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό γιατί παραλάζει την πολιτική ατζέντα η οποία απορρίφθηκε ε, στις δημοκρατικές εκλογές κάθε φορά που έγιναν δημοκρατικές εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανησυχούμε ιδιαίτερα που η παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργάνωσης υφίστανται ένα πλήγμα και είναι πρόβλημα όχι μόνο για τους ε, παραγωγούς, τους εργοστασιάρχες αλλά και για τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα σε αυτές τις μονάδες. Είναι λοιπόν μια σημαντική ανησυχία που θέλω να την πάρουν πάρα πολύ σοβαρά και να τη σκεφτούν οι συνάδελφοί μου. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για τους παραγωγούς της ΕΕ αυτή τη στιγμή γνωρίζουν μια αναπηρία σε διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο ελευθέρων συναλλαγών, εμπορίου με την πολιτική στάση η οποία υιοθετείται στην πολιτική μας ατζέντα, κάτι που τους επιβάλλεται και μου ε, ε, άκουσα τα, με προσοχή τα επιχειρήματα του κυρίου Στέρντι που μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ε, και πρέπει να το εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Συγγνώμη ε, και ένα ακόμα αίτημα. Όλοι έχουμε βοηθούς και όλοι έχουμε διάφορα πράγματα να κάνουμε. Αλλά είναι, είναι απαραίτητο να μιλάνε τόσο δυνατά οι βοηθοί μεταξύ τους μέσα στην αίθουσα. William ε, Ευχαριστώ πολύ. Άλλες παρα... παρατηρήσεις, ο κύριος Στέδη. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις συμβολές σας όλους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και είχαμε και στον Τρίλογο συζητήσεις όπως ξέρετε και βεβαίως είπαμε ναι ότι υπάρχει μια απόσυρση ε, των δασμών μας και νομίζω ότι είναι των επιστροφών ε, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε πάνω στην εισήγησή σας και στις σχετικές ε, ε, πρώτες εισηγήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πούμε ότι για το διοξίδιο του άνθρακος είναι ένα στοιχείο που γι' αυτό το λόγο το έβαλα μέσα στην έκθεση. Δεν είχαμε λάβει απόφαση όταν το έγραφα και αν παρενέβαινε η απόφαση θα ήταν πάρα πολύ αργά για να μπορέσει να δράσει η Επιτροπή και γι' αυτό το αναφέρω. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, μέγιστο και ε, αποτελεί ένα εμπόδιο στο εμπόριο και είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Δανιέλ, πρέπει να πω ότι όταν είχαμε μια συνάντηση στην ετήσια συνάντηση με όλους τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές συμφωνώ πάνω σε αυτό ότι προσπαθήσαμε να έχουμε έναν οικοδομητικό διάλογο σχετικά με την επαγρύπνηση ε, πάνω σε αυτό το θέμα ε, και βάλαμε την διατύπωση θα πρέπει και όχι θα μπορούσε κάτι το οποίο αλλάζει τον τόνο της ε, της φράσης αυτής και πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει υπόλογη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η Επιτροπή εάν δεν άλλαζε αυτά τα μέτρα. Επίσης για το ελεύθερο εμπόριο ο Βίλιαμ ε, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ότι αναπτύσσει μεγάλες ευκαιρίες και ότι πολλές φορές μπορεί να αποτελεί μειονεκτήματα για τη μία πλευρά. Όταν μιλάμε για ελεύθερο εμπόριο πρέπει να έχουν πλεονεκτήματα και οι δύο πλευρές και να υπάρχει ισοτιμία ε, και για τις δύο πλευρές. Γι' αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο το είχαμε συζητήσει και με τους άλλους σκιώδεις εισηγητές ε, όταν μιλούσαμε για αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι τίθεται εδώ ένα πρόβλημα. Υπάρχουν οι επενδύσεις των υπηρεσιών από τη μία πλευρά και εμείς έχουμε να ανταποκριθούμε σε μία πρόκληση, έχουμε μια τεράστια ευκαιρία μπροστά μας και πρέπει να την αδράξουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ισοτιμία και ότι είναι δίκαιη και για τις δύο πλευρές. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε και θα επανέλθω στην συνέχεια. Ευχαριστώ. Ε, η, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι... The files and uh, Την ε, επόμενη εβδομάδα the interim partnership agreements between the European Community. Έγινε μια συζήτηση ε, σύσταση ε, για ε, τα θέματα ανάπτυξης και συνεργασίας για το ίδιο ε, θέμα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το 2000 ε, η ΕΕ συμφώνησε για μια νέα, είχε μια νέα εμπορική ε, συμφωνία με νέους κανόνες για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος με σκοπό να γίνει μια αντικατάσταση της προηγούμενης συμφωνίας από την καινούργια σε σχέση με τις χώρες ΑΚΕ οι οποίες θα έπρεπε να υπογράψουν τη νέα ε, συμφωνία εταιρικότητας. Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για αυτή τη νέα συμφωνία το 2002 με στόχο να συμπεριληφθεί ε, το 2007 αλλά ήταν κάτι που δεν έγινε δυνατό γιατί δεν ε, υπήρξε μια συνολική συμφωνία για όλη την περιοχή, την ευρύτερη του ειρηνικού και ε, υπήρξε εστιασμός στα εμπορικά αγαθά και ε, μια δυνατότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι το πέρας του 2007 περιμένοντας μια οριστική συμφωνία για την εταιρική σχέση. Μόνο τα Φίτζι και η Παππούα ε, ε, δήλωσαν ότι θέλουν να πάρουν μέρος στις προσωρινές συμφωνίες. Με την υπάρχουσα διαδικασία έχουμε και μια προφορική ερώτηση και στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που θα ακολουθηθεί και από ένα ψήφισμα. Θα ήθελα να αρχίσουμε την συζήτηση δίνοντας το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ντέβιτ Μάρτιν από την ομάδα έρευνας και ανάπτυξης. because we had, as you, you've given a full introduction and we had a discussion on previous... Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. ε, θα ήθελα καταρχήν να ε, αναφερθώ στο σημείο 7 που αφορά το αν θα δώσουμε σύμφωνη, τη σύμφωνη γνώμη μας. Το θέμα είναι να πούμε είναι ή όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ενδιάμεσες ε, στάσεις και δυνατότητες. Ε, έχουμε συζήτηση επίσης για, τα, για τα νησιά ε, Φίτζι όπου είχαμε συζητήσει στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και για την Παπουασία ε, Τώρα το αν πούμε ναι στη συνεταιρική σχέση, στη συμφωνία περί εταιρικής σχέσης, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε επιμέρους παρατηρήσεις. Για το σημείο 7 θα ήθελα το Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του για την Παπουασία Νέα Γουινέα υπάρχουν ορισμένες επικρίσεις ε, σχετικά με αυτό το θέμα και βεβαίως ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει η προσωρινή αυτή συμφωνία ε, εταιρικότητας να επεκταθεί στα, στον τομέα της ζάχαρης και στην, σταλιευτικά προϊόντα για, που είναι προς το συμφέρον για και των δύο αυτών χωρών οι οποίες θέλουν να υπογράψουν ε, γιατί δεν θέλουν μια νέα καταστροφή στα προϊόντα του εμπορίου και στις, εταιρικ... στις εμπορικές σχέσεις. Ό,τι αφορά τώρα την αλία υπάρχει μια ανησυχία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της αλίας του τόνου από ισπανικής πλευράς και ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες ανησυχίες ε, έχω διαφορετικά συμπεράσματα προσωπικά. Πιστεύουμε ότι ε, δεν είναι δυνατόν να προκύψει ε, κάτι το οριστικό γιατί υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη ισορροπίας σε αυτή την αγορά. Η αλλαγή σε αυτή τη συμφωνία δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή αγορά αλίας. Ε, εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να απαντήσουμε στο παλαιό ερώτημα που έχουμε, στο αίτημα που έχουμε θέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραγωγή μιας ε, έκθεσης που θα αφορά την ε, διάρκεια των αλλιευτικών αποθεμάτων σε την περιοχή του Ειρηνικού ε, στο εν πάση περιπτώσει στο κοινοβούλιο θα πρέπει να παρουσιαστεί μια ε, εισήγηση που θα αφορά τις ε, την αλλιευτική συμφωνία και τις ε, εμπορικές επιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά την εμπορική ε, σε ό,τι αφορά την αλία της Ευρώπης υπάρχουν πολλά ωφέλη και δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με τον αναπτυξιακό στόχο της Ευρώπης ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να έχουμε μια θετική αντιμετώπιση για την αλληλεία μέσα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Για τα νησιά Φίτζη τώρα είναι σαφές και έγινε ακόμα πιο σαφές ε, για μένα ότι η σχετική Γενική Διεύθυνση αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα ε, γιατί υπάρχουν μεγάλα ωφέλη για τα νησιά Φίτζη ε, και ότι θα έπρεπε ε, να υπάρξει μια προσθήκη ε, για την, στον τομέα της ζάχαρης. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι πρέπει να, να συστήσουμε στα νησιά Φίτζη να επιτελέσουν σύντομη πρόοδο για να μπορέσουν να, έχουν, να εγκαταστήσουν ένα δημοκρατικό καθεστώς στα νησιά ε, και οπότε βεβαίως θα δώσουμε ε, βοήθεια στον τομέα της ζάχαρης και στήριξη στην περίπτωση αυτή. Άλλες ανησυχίες που γνωρίσαμε ήταν καταρχήν ε, για όλα τα κράτη του Ειρηνικού, την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία παραδείγματος χάρη που είναι πολύ μεγάλη εταίρη, πολύ μεγαλύτερη ε, για την Ευρώπη. Είπαμε ότι δεν θα θέλαμε να ε, συνάψουμε συμφωνίες με αυτέ τι χώρες πριν να δούμε από κοντά όλα τα προβλήματα που έχουμε με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία το θέμα της ε, ενσωμάτωσης δεν είναι ένα πρόβλημα. Το θέμα των επιδοτήσεων ε, επίσης ε, δεν αντιμετωπίζεται σε σχέση με τους γενικότερους στόχους που έχουμε και πρέπει να πούμε ότι θα είναι δύσκολη αυτή η συμφωνία για την Ευρώπη γιατί για πολλά από αυτά τα νησιά δεν υπάρχει κάποια, ε, κάποιο σοβαρό κίνητρο. Δεν έχουν σοβαρά κίνητρα γιατί δεν έχουν μεγάλο όφελος να συνάψουν συμφωνίες μαζί μας. Εν πάση περιπτώσει εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική μας για συμφωνίες εταιρικών σχέσεων και για ενσωμάτωση όλων αυτών των νησιών με όρους στήριξης ε, ε, του εμπορίου ε, υπάρχει ένα πακέτο και είπαμε και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα αναπτυξιακό πακέτο ουσιαστικό. Το θέμα είναι όμως ότι ο προϋπολογισμός και το εμπόριο ε, θα πρέπει να είναι πιο πολύ βοηθητικός για την Παπουασία Νέα Γουινέα και το, τα νησιά Φίτζη που θα πρέπει να έχουν ένα δίκαιο μερίδιο ε, στην περίπτωση αυτή και πιστεύω ότι ε, δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα υπάρξει αυτό το δίκαιο ε, μερίδιο και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε ξανά το θέμα της Παπουασίας Νέας Γουινέας και Φίτζη σε σχέση με αυτό. Σε ό,τι αφορά το ρωτοψήφισμα θα μου, ε, πραγματικά θα μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να ακούσω τις προτάσεις σας για προσθήκες και για αλλαγές. Θα ήθελα να σας πω ότι και τα δύο θέματα αυτά είναι μέσα στην ε, Συμφωνία εταιρική Σχέσης, έχουν επισυναυθεί και γι' αυτό καλό τους συναδέλφους να τα ε, συμβουλευτούν. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία προέρχονται και από την Παπουασία Νέα Γουινέα και, και από τα Φίζη και θα είμαι ευτυχής να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω σε αυτή την Επιτροπή ότι έχουμε και μια συνεισφορά, μια γνωματοποίηση από την Επιτροπή Αλίας αυτού του οίκου για τους κανόνες καταγωγής ε, σε ό,τι αφορά τα λευτικά προϊόντα. Και υπερασπίζονται ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση ό,τι αφορά τους κανόνες καταγωγής. Να δώσω τώρα το λόγο στον Κύριο Σάβα από το ΕΛΚ. ευχαριστώ. Ε, εγώ δέχομαι να αναφερόμαστε εδώ στο κείμενο σε συγκεκριμένου κανόνε καταγωγή για τα ελευτικά προϊόντα και να ζητήσουμε από την Κομισιόν στενή παρακολούθηση των διαταξιών αυτών. Επίση, ε, είμαστε ικανοποιημένοι με την δέσμευση τη Κομισιόν να παρουσιάσει μια έκθεση για τι ειδικέ πτυχέ του ελευτικού τομέα των κρατών μελών. Τώρα, θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί αυτό το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος και μάλιστα αναφέρομαι στον αρνητικό αντίκτυπο κοινωνικό και οικονομικό που έχει το μέτρο αυτό στον ε, τομέα της αλίας ε, τόνου της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης γιατί οι χώρες του Ειρηνικού θα είναι οι κυρίες χώρες που θα ωφεληθούν από αυτή την παρέκκληση και εγώ θέλω να επισημάνω εδώ ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα είναι απαραίτητο να προσθέσουμε τα ακόλουθα στοιχεία στο ψήφισμα, κύριε Μαρτίν. Καταρχήν, να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο ε, των κανόνων καταγωγής για τα ελευτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα επί του τομέα λιαστώνου. Δεύτερον, ε, να αναφέρουμε ότι η επαναφορά των κανόνων προέλευσης σε την ε, συμφωνία δεν θα υποθέτει, δεν θα αποτελεί προηγούμενο και τρίτον, να διευκρινίσουμε ότι η ε, Σύμφωνη Εταιρική Σχέση που διαπραγματευόμαστε σήμερα δεν θα περιλαμβάνει αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη για του κανόνε καταγωγή για τα μεταποιημένα προϊόντα εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η μόνη μέθοδος έτσι ώστε αφενός να εγγυθούμε την ε, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα και την του τομέα λήψης τόνους της κοινότητας αλλά και με τις ε, χώρες GSP Plus και τις λοιπές χώρες ΑΚΕ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Ευχαριστώ τον κύριο Παμπλοσάγκουα, Ρόμπερτ Στάρντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με όλα σχεδόν όσα είπε ο Ντέιβιτ. Συγχαρητήρια, Ντέιβιτ. Πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Δίκιο έχει. Θα ήθελα βέβαια να αναφέρω κάποια σημεία σε σχέση με την αλία. Αν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισαγάγει μόνο 2% ε, των ε, ψαριών σε κονσέρβα. Και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει σημαντική ε, αύξηση και τροποποίηση. Έχω μια ερώτηση. Τα Φίτζι έχουν προβλήματα με συμμόρφωση ε, με το SPS, με τα φυγειονομικά και φυτογειονομικά μέτρα. Δεν ξέρω, ίσως ο Πάμπλο να ξέρει περισσότερα σε σχέση με το γιατί ή μήπω η Κομισιό να μπορούσε να απαντήσει την ερώτηση αυτή. Κάτι άλλο για την ε, βιομηχανία της ζάχαρης. Όπως ξέρεις, εγώ εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαι με τον τομέα αυτό και πάντοτε αισθανόμουν ότι αυτό το αγαθό θα έπρεπε να την κάνει ενίσχυση, ε, κυρίως ε, για τα άτομα που βασίζονται, που έχουν εισόδημα με αυτή τη βιομηχανία. Εμείς θεωρούμε ότι όσο το συντομότερο έχουμε συμφωνία, τόσο το καλύτερο. Εγώ θα προσπαθήσω να συνεισφέρω και με την εμπειρία που έχω για αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα την Κομισιόν. Έχετε σχόλια για όσοι υπόθηκαν από τον συγητή και τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Συγγνώμη. Υπάρχει κι άλλο ένα αίτημα και θα επανέλθω στην Κομισιόν. Εργότερα ακούσουμε πρώτα τον συνάδελφο από την ομάδα Γκουα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μα... μιλήσω διαμακρών. Επανέρχομαι στις βασικές μου παρατηρήσεις ε, από την ακρόαση που κάναμε για το θέμα και με τους πρεσβευτές ε, και τους υπουργούς ε, των δύο χωρών. Ρωτώ τον εισηγητή και πάλι σε ποιο βαθμό η κοινωνική κατάσταση στις δύο χώρες εν προκειμένου λαμβάνεται υπόψη για, την, για τις περαιτέρω εξελίξεις. Ίσως ε, στην ερώτηση για προφορική απάντηση προς την Κομισιόν ε, μήπως θα έπρεπε να ρωτήσουμε σε ποιο βαθμό μια νόμιμη κυβέρνηση των νήσων Φίτζη είναι εταίρος στις διαπραγματεύσεις και εκπροσωπείται δεόντως ε, στις διαπραγματεύσεις με την Ένωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταστήσουμε σαφές με ποιον διαπραγματευόμαστε ακριβώς και τι στόχο έχουν οι διαπραγματεύσεις. Το εμπόριο και η συνεργασία θα πρέπει να γίνονται προς όφελος του πληθυσμού, του λαού των χωρών και ο λαός αυτός θα πρέπει να εκπροσωπείται νομότυπα, από νομότυπους ε, ε, εκπροσώπους. Αυτό νομίζω πρέπει να το προσθέσουμε στην προφορική ερώτηση στην Κομισιόν. Και επίσης, καλό είναι και ο εισηγητής να προχωρήσει στην υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον David Μάρτιν για την δουλειά που κάνει στα παρασκήνια για το ψήφισμα και ευχαριστώ για τις σαφείς συστάσεις σχετικά με τη διαδικασία ε, συγκατάθεσης και οι, οι φίλοι από την Παπουασία Νέου Ινέα θα συμφωνήσουν. Χαιρόμαστε για τη δουλειά που έχει γίνει από το Κοινοβούλιο στο συγκεκριμένο φάκελο. Κάποια σύντομα σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Προφανώ η ενδιάμεση συμφωνία με τι χώρε του Ειρηνικού αποτελεί μέρο μια ευρύτερη προσέγγιση με τι χώρε ΑΚΕ ε, οι μονοπλευρές ε, προτιμήσεις του Κοτονού, όπως είπατε, ε, έληξαν το 2007, όπως είπατε κι εσείς, και θα πρέπει τώρα να αναπτυχθεί μη ένα πλαίσιο προσανατολισμένο προς την ανάπτυξη στα πλαίσια του ΠΟΕ για τις χώρες του Ειρηνικού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τα σχόλια και τους όρους που έθεσε ο Ντέιβιντ σχετικά με τις δυσκολίες κάποιες από τις μικρότερες χώρες να ακολουθήσουν, εμείς συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας να, να, υπέρ των διαπραγματεύσεων για μια συνεκτική συμφωνία και υπάρχει συμφωνία ότι η συνεκτική αυτή συμφωνία θα πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ενδιάμεσης συμφωνίας, συν συνεργασία για την ανάπτυξη, ένα από τα θέματα που έθεσε ο Ντέιβιντ ένα κεφάλαιο για την αλία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και ε, διατάξεις σχετικά με την ε, σύσταση, σύνθεση. Έτσι λοιπόν ε, μιλάμε για ε, συνεκτικότητα, την οποία βέβαια ο καθένας ε, είναι ελεύθερος να την ερμηνεύει με κάπως διαφορετικό τρόπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για τη βοήθεια στο εμπόριο και τη συνεργασία εδώ γενικότερα, ο Ντέιβιντ είναι σαφής διότι ζητεί πρόσθετους πόρους. Εδώ πρέπει να κάνω μια δήλωση που είναι σημαντική. Η βοήθεια για το εμπόριο εδώ η Κομισιόν δεν μπορεί να ξεπεράσει την εντολή που έλαβε σε σχέση με το EDF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Δεν μπορεί να ξεπεράσει δηλαδή την εντολή σε σχέση με αυτές τις χώρες. Οι προσθετηπόροι θα προέρθουν από τα κράτη-μέλη ή από άλλους δωρητές. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Όμως παραμένουμε δεσμευμένοι υπέρ της ενεργού συνεργασίας με άλλους δωρητές πάνω σε αυτό το θέμα. Για να, κατα... τα καταφέρουμε θέλουμε σαφείς αξιολογήσεις από τις χώρες της περιοχής που θα εντάσσονται σε συγκεκριμένες και συνεκτικές ε, στρατηγικές ε, ελεύθερων συναλλαγών. Και η βοήθεια θα πρέπει να δίνεται μέσα από το περιφερειακό ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα τριπλασιάστηκε και τα προγράμματα που ε, υποβλήθηκαν στα πλαίσια της, στρατη... Ε, στρατηγικής σχετικά με τη βοήθεια ε, για το εμπόριο. Οπότε εδώ υπάρχει συνεργασία. Τώρα για την αλία που είναι σημαντικό θέμα, όπως αναφέρθηκε η ενδιάμεση συμφωνία περιλαμβάνει τους ειδικού κανόνες καταγωγής για προϊόντα αλληλείας, ε, Global Sourcing λέγεται, το που οδήγησε σε συζητήσεις στην Επιτροπή Αλληλείας και ετέθηκε εδώ το υπόβαθρο και οι βασικοί κανόνες εξηγούνται σε ένα κείμενο το οποίο δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες και θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η ε, Επιτροπή ε, ε, είναι υπέρ της εφαρμογής των διατάξεων Global Sourcing όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του πρωτοκόλου και αρχίζουμε διαδικασίες ελπίζουμε το 2011 να υποβληθεί σχετική έκθεση. Επίσης προβλέπεται παρόμοια διάταξη δηλαδή ε, υποβολή έκθεσης, παρακολούθηση και υποβολή έκθεσης και ε, η διατύπωση στο σχέδιο ψηφίσματος είναι Global Impact Assessment. David, αυτό είπε, σε σχέση με την συνεκτική συμφωνία στο μέλλον. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αυτά τα θέματα θα ληφθούν υπόψη δεόντως και θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη της Κομισιόν σε αυτά. Μένει μόνο ένα τελευταίο θέμα η ερώτηση του κυρίου Στέρντι. Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω σήμερα, λυπάμαι γι' αυτό. Περιορίζομαι να πω ότι τα πρότυπα SPS για φυτογειονομικά θέματα ε, θα ε, προβλέπονται. Αν υπάρξουν προβλήματα και είναι αρκετά ε, σοβαρά για να σταματήσει το εμπόριο, θα σταματήσει. Αυτό αφορά την προστασία του καταναλωτή που ενδιαφέρει όλους τους ε, ενεχομένους στη διαδικασία και υπάρχουν και ε, προγράμματα δράσης ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να ε, φάσουν στα πρότυπα αυτά. Είναι γενικά αυτά που σας λέω. Αν θέλετε κάτι πιο συγκεκριμένο θα το ψάξουμε με τους συναδέλφους από το αρμόδιο τμήμα Γενική Διεύθυνση. Νομίζω ότι κάλυψα τα σημαντικότερα θέματα. Αν υπάρχουν, και κάτι, αν υπάρχουν πιο ειδικέ ε, παρατηρήσεις, ε, μπορώ να σας παραπέμψω ή να το ψάξω. Ας επανέλθουμε στον κύριο David Μάρτιν για τελικά σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, νομίζω ότι εν γέννη συμφωνούμε Έχουμε παρόμοια προσέγγιση για το θέμα αυτό. Για τον κύριο Ζάλμπα, σας ευχαριστώ για τα επικοδομητικά σας σχόλια. Κατανοώ ότι ε, έχετε και τα δικά σας συμφέροντα από την πλευρά της Ισπανίας ε, γιατί η Ισπανική βιομηχανία είναι ιδιαίτερα εμπλεκόμενη στο θέμα αυτό αλλά μίλησα ε, και με του ε, τους και από ό,τι κατάλαβα δεν θα έχει σημαντική επίπτωση η συμφωνία αυτή τώρα ε, αλλά πρέπει να παρακολουθήσουμε και την βιωσιμότητα της ελευτικής δραστηριότητας ε, και φυσικά στο μέλλον, ε, αν ε, δούμε, παραδείγματο χάρη, μαζικά ο Κινέζικο τόλο να εμφανιστεί στην περιοχή και να έχουμε υπεραλήψη και μεταποίηση ελευτικών προϊόντων, θα επανέλθουμε στο θέμα. Αλλά αν έχετε φυσικά συγκεκριμένε τροπολογίε, ευχαρίστω να τι εξετάσω για να δούμε αν μπορούμε να τι θετήσουμε στο ψήφισμα. είπε ο Ρόμπερτ, ε, Ναι, ε, συζητήθηκαν αυτά τα θέματα μεταξύ μας και από ό,τι φαίνεται είναι τεχνικά το πρόβλημα ότι το Φίτζι μέχρι τώρα τα, τα νησιά Φίτζι δεν έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες διαδικασίες ε, για τα υγειονομικά και τα φυτογειονομικά. Ε, Φυσικά, αν ε, δεν πληρούνται αυτά τα πρότυπα, δεν θα υπάρξουν και εισαγωγέ. Ε, για όσο είπατε για τη ζάχαρη, ε, αυτό συνδέεται και με το σχόλιο του κ. Σούλτ. Αν θέλετε, για να προστατεύσουμε την συνέχιση του εμπορίου μεταξύ των νησιών Φίτζη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς κυρώσεις, ε, να σας πω ότι δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα τίποτα εκτεταμένο με τα νησιά Φίτζη και πολύ καλό παραδείγμα αποτελούν οι πόροι για τη βιομηχανία Τσάγκαρη. Σίγουρα χρειάζονται τα νησιά Φίτζη τα χρήματα αυτά, αλλά δεν θα ήταν αποδεκτό για μας ε, να χορηγήσουμε αυτά τα χρήματα αν υπάρχει στρατιωτικό πραξικόπημα στο Φίτζι, ε, ε, στα νησιά Φίτζη. Έτσι λοιπόν συμφωνούμε ότι πρέπει να το δούμε αυτό στα πλαίσια της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, όμως η Κομισιόν δεν έχει απελευθερώσει τους πόρους. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα αποκατασταθεί η δημοκρατία στα νήσου Φίτζη. Νομίζω ότι εδώ προσπαθούμε να ξεβρούμε τη σωστή ισορροπία. Λαμβάνουμε υπόψη την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Πρόεδρε, βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά αφού δεν τα θέσαμε στην αρχή, δεν νομίζω ότι είναι σωστό τώρα να τα θέσουμε στο τέλο τη συζήτηση. Από ό,τι βλέπω, διαγράφεται μια συνένεση και θα ήταν καλό να κλείσουμε εδώ το ζήτημα να επιτρέψετε μου να επιτρέψετε ότι οι τροπολογίες θα κατευθούν μέχρι τις 11 του μήνα, προθεσμία 11 Νοεμβρίου. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. τροποποίηση τη συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Αφρική για το εμπόριο την άπτυξη για τη συνεργασία Νικόλο Ρινάλντι, Άλντε, από τους φιλελεύθερους είναι ο εισηγητής. Απλώς να σας ε, υπενθυμίσω ότι η Νότια Αφρική είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος μας στην Αφρική και ε, να σας πω ότι έχουμε και τις συμφωνίες, συμφων... τις εμπορικές συμφωνίες και τις συμφωνίες εμπορική συνεργασία. Έχουμε τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών που υπεγράφει στην Πρωτορία το 1999 και τέθηκε σε ισχύ το 2004. Επομένως, καθώς ε, ε, τότε, μάλλον, ε, τότε είχαμε αποτυχία και εδώ ε, εμπίπτουν αυτές οι αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ανάπτυξης, γιατί τότε δεν υπήρχε Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Η δική μας Επιτροπή ε, οργάνωσε αποστολή στην Νότια Αφρική πρόσφατα. Ήταν πολύ χρήσιμη η επίσκεψη αυτή. Βελτιώθηκε η κατανόηση της Επιτροπής μας. Ε, σε σχέση με το πώς κινούνται τα πράγματα σε αυτή την ταχύως αναπτυσσόμενη χώρα, η οποία διδραματίζει έναν όλο ένα και πιο σημαντικό ρόλο στις ε, συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις των ΠΟΕΣ, στις συνεχιζόμενες συζητήσεις των ε, γύρω στον ΠΟΕ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Νικολό Ρινάλντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω υπενθυμίσατε και εσεί σωστά, η συμφωνία ενσυσχύει από το 2004. Είναι μια συμφωνία που συνολικά λειτουργήσε επιτυχώ. Ε, η Νότια Αφρική είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος μας ε, ε, στην Αφρική αλλά και για την Νότια Αφρική η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος. Έχουμε 34% εξαγωγές από την Νότια Αφρική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 35% αντίστροφη ροή εμπορίου. Ε, είναι πολύ στερεά η συμφωνία, σταθερή συμφωνία αυτή και απελευθέρωσε το εμπόριο σχεδόν όλων των προϊόντων μεταξύ ε, των ε, δύο εταίρων μέσω και ενός μηχανισμού γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων για κάποια προϊόντα. Υπάρχουν βέβαια κάποιε εξαιρέσει για πολύ ευαίσθητου τομεί, ορισμένα αγροτικά προϊόντα από την Νότια Αφρική και ε, ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα από την πλευρά της Ευρώπης όπως ε, η φαντουργία και η διένδυση. Το 2005 το Κοινό Συμβούλιο Συνεργασίας υιοθέτησε μια σειρά τροπολογιών. Δεν έχω πολλά να πω από αυτόν γιατί ε, έχουμε παρόμοιες τροπολογίες στη συμφωνία αλλά κυρίως πρόκειται για γλωσσικές τροπολογίες απλώς βελτιώνουν ορισμένα τμήματα της συμφωνίας. Εκεί όπου μιλάμε για δίκτυα μεταφορών, θέλαμε να προσθέσουμε ότι πρόκειται για ασφαλές δίκτυα μεταφορών. Εκεί όπου μιλάμε για συνεργασία, για την ενίσχυση της ασφάλειας, της αερομεταφορές, ε, μιλάμε ε, και για αερομεταφορές, αλλά και για σιδηροδρομικές μεταφορές. Εκεί όπου μιλάμε για ε, ασφάλεια και υγεία, βάλαμε, προσθέσαμε και προστασία του περιβάλλοντος, ασφάλεια περιβαλλοντική κτλ και από την πρόταση χρηματοδότηση περνάμε στο σχέδιο, ετήσιο σχέδιο δράση που εκπονήθηκε. Έτσι λοιπόν πρόκειται για μια σειρά τροπολογιών τεχνικού χαρακτήρα επί τη ουσία που δεν ε, χρειάζεται ε, να τις αξιολογήσουμε πολιτικά. Η γνωμοδότηση ε, που δίνουμε τώρα εμείς στην Επιτροπή Ανάπτυξης είναι να αναφερθεί στην ανάπτυξη της δικής μας πολιτικής εναντί της Νοτιού Αφρικής. Είναι μια χώρα που επισκεφθήκαμε εμείς προ λίγων ημερών Είχαμε την επιβεβαίωση των όσων γνωρίζουμε ήδη. Υπάρχουν ε, ε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αντικειμενικά στοιχεία. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική από οικονομική και εμπορική σκοπιά στη χώρα αυτή, αλλά θα έλεγα ότι κυρίως ίσως ε, θα έπρεπε να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για μια χώρα η οποία είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη ψυχολογικά, από ψυχολογική σκοπιά, δηλαδή και για το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει στην ευρύτερη ε, μεσημβρινή Αφρική, αλλά και σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο. Ε, οργανώνεται και έχει φιλοδοξίες προκειμένου να γίνει μια πραγματική υπερδύναμη σε περιφερειακό επίπεδο. Αλλά πρόκειται και μια πολύ φιλόδοξη χώρα και στα πλαίσια του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων που διεξάγει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν έχει ξεκαθαρίσει ιδέες και απόψεις και επιζητά να πουλήσει τη θέση της ε, στην πιο ακριβή τιμή αν θέλετε. Επίσης πρόκειται για μια χώρα ε, στην οποία λαμβάνει μια πραγματική, χώρα μια πραγματική εσωτερική συζήτηση σε σχέση με άλλες αφρικανικές χώρες. Μάλιστα βλέπουμε και ποικιλή απόψεων ορισμένων θεμάτων και όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στις τροπολογίες που έγιναν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ε, από την πλευρά των Νότιοφρικανών για τη συμφωνία αυτή. Ίσονο σημασία, επαναλαμβάνω, αλλά μας επιβεβαιώνουν ότι προσέχουν πάρα πολύ τις λεπτομέρειες, ότι θέλουν να εξειδικεύσουν μια σειρά προβληματικών, δεν αφήσουν τίποτα στην τύχη και επομένως είναι ιδιαίτερα σχολαστική. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε ε, σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψε να δώσουμε μία έγκριση και στις τροπολογίες αλλά ε, και στην ε, γνωμοδότηση, την αιτιολογική έκθεση που στέλνουμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης όπου τοποθετούμαστε σε σχέση με την εξέλιξη των σχέσεων μας με την Νότια Αφρική. Τώρα, τι θα κάνουμε εμείς με την Νότια Αφρική επί πτυχών. Εδώ θα βασιστούμε ίσως σε κάποιες εμπειρίες ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και θα μπορούσαμε να τις εφαρμόσουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Ε, πρέπει συνεχώς να επικαιρώνουμε τη συμφωνία που έχουμε και από τη σκοπιά της ορολογίας Έχουμε λοιπόν κάποιου συνομιλητέ που είναι απαιτητικοί και τι συμβαίνει με την Νότια Αφρική. Εγώ νομίζω ότι αυτή θα είναι μια εμπειρία που μπορεί να είναι χρήσιμη και με άλλε δυνάμει όπω Βραζιλία, Ινδία, αναπτυσσόμενε χώρε ε, δηλαδή, ε, όπου ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, 40% είναι κάτω από το όριο τη φτώχεια, αλλά υπάρχει παρόλα αυτά δυναμική και έχουν και δυνατότητε οικονομική αριστεία. Εγώ δυστυχώ ε, σήμερα δεν θα είμαι παρόν, σήμερα το απόγευμα. Ε, στη συζήτηση για την ε, ε, εταιρική σχέση για τις χώρες ΚΑΜΑ, για την κοινότητα για την ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής. Έχουμε υποδιαπραγμάτευση μια συμφωνία εταιρική σχέσης και με την κοινότητα αυτή. Υποδιαπραγμάτευση Τώρα θέλω να κλείσω την παρουσίασή μου με μια σκέψη που εκφράσαμε ε, στην Νότια Αφρική κατά την επισκέψη της αντιπροσωπείας. Ίσως ε, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε είτε ως πολιτικές ομάδες είτε ως Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να κάνουμε μια συζήτηση στην Ελλομέλεια πριν τα τέλη του έτους επί της πολιτικής ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτιού Αφρικής ε, εν ώψη της ε, ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με την Νότια Αφρική για την UNAB. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θα μας επιτρέψει να εξορθολογήσουμε αυτές τις εμπορικές σχέσεις στις οποίες ε, αναφέρεται τώρα η δική μου έκθεση και οι τροπολογίες. Ευχαριστούμε, Νικολινάλντι. Θέλουν ε, κάποιοι να συμμετέχουν στη συζήτηση. Θέλει κάποιος το λόγο. Αλλιώς θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Κάρλος Βερμέχο. Where is the Okay, Όχι. Από την Κομισιόν δεν υπάρχει κανείς για να μιλήσει. Άλλος από την Επιτροπή, ο κύριος Λάγκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η διεύρυνση της εμπορική συμφωνίας με την Νότια Αφρική είναι επίκαιρο θέμα και απαραίτητη. Το 1994 αρχίσαμε, μετά το τέλος της Apartheid, αρχίσαμε τι διαπραγματεύσει με την Νότια Αφρική και τότε ήταν πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν τέσσερα χρόνια. Γιατί υπήρχαν πολλά επιμέρους που προσέκρουαν σε αντιδράσει των κρατών μελών και έτσι η εταιρική ανταλλαγή δεν προχωρούσε τόσο γρήγορα όσο είχαμε φανταστεί. Γι' αυτό χαιρετίζω τη νέα αυτή εκκίνηση, αλλά σε αυτό το θέμα είναι σημαντικό να πιάσουμε και ευαίσθητους τομείς. Ε, λεπτά θέματα ευαίσθητα κυρίως για την Ευρώπη, αλλά και προοπτικές ανάπτυξης, που συνεπάγονται προοπτικές ανάπτυξης για την Νότιο Αφρική. Στον τομέα της ζάχαρης, για παράδειγμα, που ιδιαίτερα στον τομέα του empowering αναπτύσσει νέες δυνατότητες και παίζει μεγάλο ρόλο για τον ε, κόσμο στη Νότια Αφρική. Γι' αυτό χρειάζεται εδώ να βελτιώσουμε τις συνθήκες πρόσβασης στην αγορά. Ναι λοιπόν, στο να καταπιαστούμε με αυτό το θέμα, αλλά να το διαμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψει από εδώ μια εταιρική σχέση. Ευχαριστούμε. Άλλα σχόλια, ο Νικολά Ρινάλντι έχει να σχολιάσει. Μια παρατήρηση να επαναλάβω η δική μου έκθεση αποτελεί την ευκαιρία να προβληματιστούμε επί της πολιτικής που ακολουθούμε έναντι της Νοτιού Όμως δεν πρέπει να εμπλέξουμε για τα διάφορα ζητήματα σε σχέση με τη Συμφωνία εταιρική Σχέσης για την Νοτιοαφρική γιατί αυτά είναι ξεχωριστά ζητήματα. Πρέπει να το εξετάσουμε ξεχωριστά αυτό το θέμα. Όμως επαναλαμβάνω ότι για ορισμένες πτυχές, ακόμη και ορισμένα θέματα που αφορούν αυτές τις ε, τροπολογίες και ε, κυρίως οι διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα στην Πρωτορία και στις Βρυξέλλες. Για όλα αυτά θα είναι σκόπιμο να κάνουμε μια συζήτηση στην Ολομέλεια όπου θα αξιολογηθεί και το έργο που θα έχει γίνει από την αντιπροσωπεία μας τις προηγούμενες ημέρες. Yes, uh, let me remind you that the consideration of draft opinion will take place. Λοιπόν, θα εξεταστεί το σχέδιο γνωμοδότης στη συνεδρίασή μας, ε, στη συνεδρίαση που θα έχουμε 1 και 2 Δεκεμβρίου φέτος. Και έτσι τελειώσαμε και αυτό το θέμα. So we are we are expecting the arrival of Commissioner De Gucht. Λοιπόν, ο Επίτροπος Δεγκούχτ. Έχει σειρά τώρα. Α, δεν ήρθα ακόμα. Α, ε, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Να αρχίσουμε το σημείο 10, συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδίας, Λίχτενστάιν και Νορβηγίας. Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλληλείας. Εκλήθη το Κοινοβούλιο να εξετάσει το πακέτο αυτών των συμφωνιών μεταξύ Ένωσης και αυτών των τριών χωρών για τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 2009-2014 και τα πρωτόκολλα για τα, τις ε, παραχωρήσεις ε, ε, στην ε, Ισλανδία και την Νορβηγία. Η Επιτροπή Ελίας ήδη έχει εγκρίνει τη γνωμοδότησή της στην έκθεση αυτή και συστήνει στο Κοινοβούλιο να συγκατατεθεί στις συμφωνίες. Εμείς είμαστε η καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή και η συγγήτριά μας είναι η κυρία Μαρία Ελένη Κόπα από την ε, Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και της δίνει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον ε, περασμένο Δεκέμβρη το Συμβούλιο ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για να συνεχίσει να ισχύει η συμφωνία που είχε ξεκινήσει το 1994 ανάμεσα στα κράτη-μέλη που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή αφορά τα ποσά που καταβάλουν η Ισλανδία, το Λίχτενστάιν και η Νορβηγία ως αντιστάθμισμα και τα οποία συμβάλλουν στην άβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Η περίοδος είναι κάθε φορά πενταετής. Η τελευταία περίοδος χρηματοδοτικής συνεισφοράς έληξε το 2009 για την επόμενη περίοδο 2009-2014 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις το Σεπτέμβριο του 2008. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων παρουσιάστηκαν δυσκολίες που είχαν να κάνουν με την αύξηση που ζήτησε το Συμβούλιο στα κονδύλια για τον νορβηγικό χρηματοδοτικό μηχανισμό. Το τελικό κείμενο, όπως είπατε, περιλαμβάνει τέσσερες συμφωνίες που παρέχουν ένα συνολικό πακέτο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το οποίο αποτελείται από αύξηση 31% του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και από αύξηση 22% του νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν στις 12 πιο νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Οι τομείς προτεραιότητες προτεραιότητας όπου θα διοχετευτούν οι χρηματοδοτικές συνεισφορές είναι η προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κοινωνία των πολιτών, η κοινωνική ανάπτυξη και τέλος η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Συμφωνία παρέχει τη δυνατότητα επανεξέτασης τον Νοέμβρη του 2011 και τον Νοέμβρη του 2013 με σκοπό την επανεκτίμηση τυχών μη δεσμευθέντων διαθέσιμων κεφαλαίων. Γέργα μεγάλης προτεραιότητας για τα δικαιούχα κράτη. Η συμφωνία που επετεύχθη σε επίπεδο Συμβουλίου εκφράζει, θεωρώ, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προτείνω την έγκρισή της. Commission. Let's, uh, thank you. Let's listen to the Commission. Θα ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαρτίνα Ρέιμαν ή ο Πίτερ Μάιερ. Ποιος θα πάρει το λόγο. Ο κύριος Πίτερ Μάιερ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι ο Πίτερ Μάγερ, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν ε, για αυτήν την πολύ θετική εισήγηση την οποία εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος και ε, θα ήθελα να θε, θεωρώ ότι δεν θέλω να χάσουμε χρόνο, δεν είναι καλό να χάσουμε χρόνο με ειδικέ ερωτήσεις και θέματα. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις, την αύξηση των ε, ε, οικονομικών ε, στηρίξεων και να δούμε γενικά τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε αυτούς τους μηχανισμούς ε, σύμφωνα με τις πρακτικές της ΕΕ. Αυτά τα προγράμματα κατά προσέγγιση τα οποία ε, πιστεύουμε ότι θα δώσουν μεγαλύτερη συνεκτικότητα και ο περισσότερο όφελος σε όλες αυτές τις ε, χώρες που παίρνουν μέρος στις συμφωνίες με την ΕΕ. Ευχαριστώ πολύ άλλα μέλη της Επιτροπής ίσως θέλουν να λάβουν το λόγο. Δεν θέλει κανείς να λάβει το λόγο. Ε, η Μαρία Ελένη, εάν συμφωνούν οι σκιώδεις εισηγητές με αυτά θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ε, περαιτέρω ε, με τη σύσταση. Να συμφωνήσουμε δηλαδή πάμε με την έγκριση του σχεδίου σύστασης. Ωραία, λέει ο Προεδρεύων. Τελειώσαμε με το 10 και ε, τώρα ε, ήρθε ο Επίτροπος Δεγκούχ, τον οποίο καλωσορίζω. Μόλις έφτασε στην Επιτροπή μας. Ο στόχος ε, της ανταλλαγής απόψεων με τον Κάρελ Ντεγκούχ, τον αρμόδιο επίτροπο, είναι να έχουμε μια γενικότερη παρουσίαση των ε, ε, συμφωνιών περί ε, εμπορικής πολιτικής. Είναι η καινούρια συμφωνία για την αύξηση του εμπορίου και για, τις, ε, για τα κύρια σημεία της ευρωπαϊκής στρατηγικής από ε, αυτής της ε, συμφωνίας. Θέλουμε δηλαδή να δούμε τα διάφορα εμπορικά σημεία, τα σημεία που αφορούν το εμπόριο σε σχέση με αυτή τη συμφωνία την οποία διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι είναι μια νέα θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία πιστεύει με ότι με μια σωστή εμπορική συμφωνία θα μπορούσε, θα μπορέσει μάλλον να έχει καλύτερες, ε, μια καλύτερη στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ανάπτυξης ε, περιβάλλοντος και θέλουμε να συζητήσουμε αυτήν την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά όταν συζητήσαμε την έκθεση του κυρίου Γκάσπαρη πάνω σε αυτό το θέμα είδαμε πόσο ενδιαφέρον υπήρξε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ντεγκούχ, το οποίο έλαβε την απόφαση να έρθει στην Επιτροπή μας για να παρουσιάσει για πρώτη φορά, και αυτό έχει συμβολική αξία, αυτή τη συμφωνία στην Επιτροπή μας. Είναι ο πρώτος δημόσιος λόγος που εκφωνεί πάνω σε αυτό το θέμα, που αφορά όλες τις ε, αλλαγές ε, και η συνθήκη της Λισαβόνας επέφερε πάρα πολλές ε, αλλαγές στις σχέσεις Επιτροπής και Κοινοβουλίου πάνω σε θέματα εμπορίου. Έχουμε μισή ώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε, χωρίς να χρονοτριβήσουμε θα ήθελα να σας δώσω το λόγο και μετά που θα έχετε περατώσει την ομιλία σας θα δώσω τουλάχιστον το λόγο σε ένα μέλος της Επιτροπής μας που θα μιλήσει σχετικά με την ανακοίνωσή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη λίγα λεπτά πριν μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημα ενέκρινε αυτή τη νέα στρατηγική για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τις παγκόσμιες υποθέσεις. Είναι ένα καυτό θέμα που βγαίνει από το φούρνο. Μόλις τώρα ε, δίνεται, ε, δόθηκε στα, ε, στον τύπο και σήμερα θα ήθελα να σας δώσω μια πρώτη γεύση αυτού του θέματος μέσα από την ανακοίνωσή μου. Θα ήθελα να σας πω ότι βεβαίως υπάρχει κάποια επιφύλαξη επιφύλαξη γιατί δεν είχατε την ε, ευκαιρία να διαβάσετε αυτό το κείμενο για να μπορέσετε να αντιδράσετε σωστά. Θα έχουμε αργότερα λοιπόν τις ε, αντιδράσεις σας. Αργότερα θα έχουμε ε, ανακοίνωση στο, στα ΜΜΕ και αύριο το βράδυ θα συναντήσω τους Υπουργούς Εμπορίου της ΕΕ για να παρουσιάσω αυτή την ανακοίνωση και σε εκείνους. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση η οποία οποία είναι αποτέλεσμα μιας δημόσιας διαβούλευσης 300 σχόλια και παραπάνω, μια γενική επισκόπηση με το Ευρωβαρόμετρο υπήρξε για τα 27 κράτη-μέλη σε σχέση με τη στάση τους ως προς το εμπόριο. Η εφετηρία για την, αυτή την ανακοίνωση είναι η αναγνώριση ότι η Ευρώπη πάντοτε είχε προβλήματα σε σχέση με το εμπόριο και βεβαίως ε, αυτά υπήρχαν γιατί η Ευρώπη θέλει να πετύχει έναν υψηλό στόχο. Δεν είναι αυτό σκοπός το εμπόριο για την Ευρώπη. Πρέπει να πούμε επίσης ότι 60 χρόνια σχεδόν μετά από την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αλλάξει οι πολιτικές και κυριότερα η ε, περιφερειακή ενσωμάτωση και ολοκλήρωση. Ε, εξωτερικά πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι οι φτωχότερες χώρες του κόσμου εισέρχονται σε αυτό το πλαίσιο ε, που δεν έχει δασμούς, που δεν έχει ποσοστώσεις και δίδονται και οι σωστές βάσεις για τα ε, δικαιώματα τα εργασιακά και τις συνθήκες εργασίας. Είναι πολύ βασικό αυτό και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και για τους εργαζομένους και είναι καλό και για τους ανθρώπους και για τις χώρες στον κόσμο ολόκληρο. Αυτή η ανανεωμένη εμπορική πολιτική στηρίζεται στις επιτυχίες της ε, ε, Καθολικής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2006 και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση που αναλάβαμε να διεκπαιρεώσουμε όλες τις συμφωνίες ε, τις εμπορικές οι οποίες ε, παρουσιάζουν εκκρεμότητες και δεν προσπαθούμε να βεβαίως να εφεύρουμε εκ νέου τον τροχό αλλά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα γιατί μετακινήθηκε η πολιτική μας από το 2006 και πρέπει να αντικατοπτρίσουμε αυτές τις αλλαγές στην καινούρια μας πολιτική. Καταρχήν ε, διανύουμε μια οικονομική κρίση και πρέπει να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας ούτω ώστε το εμπόριο να έχει περισσότερη παροχή εργασίας και περισσότερη αύξηση μέσα στα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση, να εξέλθουμε από αυτήν και αυτό το βλέπουμε και στον υπότιτλο της ανακοίνωσής μας, εμπορευματική πολιτική σαν ένα στοιχείο ε, θεμελιακό για την στρατηγική του 2020 της ΕΕ. Δεύτερον, η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει ένα νεοθεσμικό πλαίσιο και με όρους εύρους της ε, εμπορικής πολιτικής και με όρους του πώς θέλουμε να δώσουμε το μήνυμά μας σχετικά με αυτή την πολιτική. Καταρχήν υπάρχει μια νέα στρατηγική, το Κοινοβούλιο έχει αυξημένες ε, δικαιοδοσίες, αυξημένο ρόλο στον ε, εμπορικό τομέα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντική αλλαγή. Καταρχήν δουλεύει πολύ σωστά. Έχουμε ε, τους, τις, ε, τα θέματα της ε, Νότιας Κορέας, τα, τα, θέματα των Δυτικών Βαλκανίων και ένα διάστημα που διανύεται ανάμεσα στα δύο είναι και το θέμα των, της δράσης γενικότερα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα έξι σημεία να τονίσω για την ανανέωση της πολιτικής μας. Καταρχήν πρέπει να είμαστε σοβαροί για να περατώσουμε αυτά που έχουμε ήδη υποσχεθεί. Ε, μετά από τον γύρο της Ντόχα, μετά από διμερείς συμφωνίες θα αναπτύξουμε ε, σχέσεις εταιρικές με διάφορα σημεία του κόσμου και θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Ε, χρειάζεται να έχουμε μια ε, πολύ σωστή ανάληψη ευθυνών και θα πρέπει να είναι σωστός διαπραγματευτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εσείς και το Συμβούλιο θα διαδραματίσετε ένα πολύ σοβαρό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε ιστορία κοινή με το Κοινοβούλιο και γι' αυτό ε, έχετε την σωστή πληροφόρηση σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων ούτως ώστε να μπορείτε να διαδραματίσετε έναν επίσημο ρόλο ε, μέσα στη διαδικασία. Ύστερα θα πρέπει να εμβαθύνουμε τις ε, σχέσεις μας ως προς τις επενδύσεις και το εμπόριο και με άλλους μεγάλους εταίρους, τις Ηνωμένε Πολιτείε, την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Ρωσία και να οικοδομήσουμε σωστά τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πάνω σε στρατογικές εταιρικότητες. Ε, υπάρχει και το θέμα της κατάργησης των ε, δασμών για το εμπόριο και τις ε, επενδύσεις. Χρειαζόμαστε για την ώρα ένα διάλογο με την Κίνα υψηλού επίπεδου και να καθορίσουμε τις οικονομικές σχέσεις μας με όλες αυτές τις χώρες και να προβλέψουμε για το μέλλον και να επιλύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν ή που πρόκειται να υπάρξουν, τα τρέχοντα προβλήματα αλλά και τα μελλοντικά. Αυτά τα φόρμ θα συναντηθούν το Δεκέμβριο και τα δύο και πρέπει να δούμε υπό το φως όλων αυτών το πόσο θα σχηματίσουμε τις καινούριε μας σχέσεις με άλλους εταίρους κλειδιά. Ε, τα θέματα τα συνολικά του εμπορίου εξελίσσονται επίσης γιατί υπάρχει ανταπόκριση των, η περικοπή των δασμών είναι ε, μία άρση των εμποδίων κάτι το οποίο σημαίνει άρση των ρυθμιστικών εμποδίων, οπότε έχουμε καλύτερες επενδύσεις, έχουμε άνοιγμα των δημοσίων προμηθειών, καλύτερη προστασία της ε, ε, πνευματικής ιδιοκτησίας ε, και στα θέματα των πρώτων υλών και της ενέργειας επίσης καλύτερη προμήθευση. Έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη στα θέματα της εμπορικής ατζέντα μας. Μέχρι το 2020 πρέπει να υψωθούμε σε ένα επίπεδο ΑΕΠ της ΕΕ που να ξεπερνάει το 1%, να είναι 1% ψηλότερο από ό,τι θα ήταν διαφορετικά. Πρέπει επίσης να έχουμε εσωτερική ανάπτυξη, κινητοποίηση για την αύξηση και για τις θέσεις εργασίας. Ε, έτσι η παγκοσμιοποίηση ε, δεν κάνει πια διακρίσεις ανάμεσα στις πολιτικές που αφορούν το εσωτερικό και το εξωτερικό της ΕΕ. Έχουμε ε, συνολικές καθολικές αγορές και το πρόβλημα είναι η πρόσβασή μας σε αυτές ανεξαρτήτως μεγέθους. Ε, η νέα εξωτερική υπηρεσία θα πρέπει να έχει έναν πολύ σοβαρό ρόλο σε όλα αυτά και επίσης ε, θέλουμε πρόσβαση στις αγορές των εταίρων μας και όπως και αυτές οι χώρες θα πρέπει να έχουν μια σωστή απολαβή των δημοσίων ευρωπαϊκών αγορών της ΕΕ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ασυμμετρία σε αυτές τις διαδικασίες αλλά ανοιχτό χαρακτήρας. Ε, πρέπει να πούμε ότι πάνω από 4,6% εκατομμύρια ανθρώπων δουλεύουν για εταιρείε αμερικανικές και ιαπωνικές μέσα στην ΕΕ μόνο. Θέλω λοιπόν να υπάρξουν μέτρα ε, πλήρη για τις επενδύσεις, τις εμπορικές με τους εταίρους κλειδιά. Αυτό είναι επίγον, ειδικά για χώρες όπως η Ινδία, ο Καναδάς και η Σιγκαπούρη, όπου οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά. Επίσης θέλουμε να δούμε το ενδεχόμενο μια αύξηση τη ευθύνη τη ΕΕ για διεθνεί επενδύσει. Αυτό που πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Πέμπτον, προτείνω να έχουμε μία πιο τολμηρή προσέγγιση στην ενίσχυση των εμπορικών συμφωνιών για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι κανόνες εφαρμόζονται ισότιμα για όλους. Θέλουμε να διασφαλίσουμε το γεγονός ότι η εμπορευματική πολιτική μας ε, αποφέρει ωφέλη. Ο στόχος μας είναι όχι να υπογράψουμε συμφωνίες απλώς, αλλά να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ένα πλήρες δυναμικό ανάπτυξης αυτών των συμφωνιών ε, και ότι χρειάζονται όλες αυτές ενίσχυση. Ε, απορρίπτει η Ευρώπη τον προστατευτισμό και τελικά θέλει να είναι σίγουρη ότι οι πάντες εποφελούνται από τα ωφέλη της καθολικής οικονομίας. Αυτό εφαρμόζεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολύ περισσότερο στον αναπτυσσόμενο κόσμο όπου το εμπόριο πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν μια χείρα βοηθείας την οικονομική πρόοδο και την ε, ενσωμάτωση στην περιφερειακή αγορά και αγορά εργασίας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι για, τα επόμενα, για το επόμενο έτος υπάρχουν ορισμένες αναμονές για την εμπορική πολιτική, η οποία πρέπει να προωθηθεί. Πρώτον, πρέπει να δουλέψουμε για μια σύναψη συμφωνίας ε, πρόορη ε, ε, για, με την Τόχα. Πιστεύουμε ότι θα, η συνάντηση κορυφής του G20 θα δώσει μια νέα όθηση για να περατώσουμε τη συμφωνία αυτή μέσα στο 2011 και θα υπάρξει μια αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πάει στη Γενέβη για μια υπουργική συνάντηση. Δεύτερον, ε, πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε πέρα από την Τόχα. Θα υπάρξει ε, μια ομάδα προσωπικότητων από αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες για να συντάξουν την άποψη της Ευρώπης για την μελλοντική κατεύθυνση και τη λειτουργία του ΠΟΕ μετά από την Τόχα. Αυτό θα γίνει μέσα στο 2011 12. Τρίτον, διμερός θα πρέπει να έχουμε άκτα για τις συμφωνίες με την ε, Νότια Κορέα και στο τέλος του επόμενου έτους με την Κεντρική Αφρική, το Περού και την Κολομβία. Σε αυτή τη φάση θα έχουμε επίσης συμφωνίες με την Ινδία, τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη, την Ουκρανία και το Μερκοσούρ. Όλα αυτά είναι δύσκολα θέματα αλλά, ε, γιατί είναι πολιτικά ευαίσθητα αλλά θα πρέπει να περατωθούν οι συμφωνίες αυτές μέσα στο 2011. Θα θέλαμε να έχουμε ε, επίσης ε, καλύτερες διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας στον, ε, στην Ένωση Νότιο-Ανατολικών Ασιατικών Εθνών όπως είναι η Μαλαισία και το Βιετνάμ. Τέταρτον, ο Επίτροπος Μπαρνιέ και εγώ θα προχωρήσουμε στο δεύτερο ήμιση του φετινού έτους στην εκπόνηση νέων ιδεών για, να το, για τη διασφάλιση της, των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών και της συνεργασίας, της υποστήριξης του εμπορίου και των ανοιχτών αγορών. Πέμπτον, θα προτείνουμε αναδιάρθρωση του γενικού συστήματος προτιμήσεων για τις αναπτυσσόμενες χώρες και θα υπάρξει μια ανακοίνωση της Επιτροπής για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Έτσι, στη συνέχεια θα έχουμε σύναψη οικονομικών συμφωνιών εταιρικότητας με αφρικανικές χώρες και χώρες του ειρηνικού. Θα παρουσιάσουμε έκτον δύο περαιτέρω ε, πρωτοβουλίες, μία πράσινη για βελτίωση ε, ε, του συστήματος εξαγωγών μας γιατί υπάρχει το θέμα ε, των περικοπών σε ορισμένους ευαίσθητους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας και στη συνέχεια θα γίνει μια ανακοίνωση από τον Αντιπρόεδρο Ταζάνη για, τις, για τα μέτρα στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μο, πρέ, πρέπει να προαχθούν γιατί μόνο ένα από τα 7 ε, κράτη-μέλη έχει δραστήριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ύστερα θα πρέπει να παράγουμε μια ετήσια εισήγηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση με τα εμπόδια του εμπορίου και, της, και των επενδύσεων. Εμείς και εννοώ και εμείς και η Επιτροπή σας αλλά και εγώ θα είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι μέσα στο 2011 πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Θα συνεργαστούμε Ευχαριστούμε από, με την Επιτροπή σας πάρα πολύ στενά. Είστε οι πρώτοι που πληροφορούμε και ελπίζω να ακούσω τώρα τις πρώτες αντιδράσεις σας και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σε μια επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, έχετε πάρα πολλά θέματα στην για διάταξη για τα επόμενα χρόνια. Όπως σας είπα, είχαμε ως στόχο να ακούσουμε τον Επίτροπο να μας παρουσιάσει αυτή την ε, πολιτική που θα ακολουθήσει η Κομισιόν. Δεν είχαμε σκοπό να κάνουμε μια πλήρη συζήτηση για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, το επόμενο τέταρτο, για να έχουμε κάποιες αντιδράσεις. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν επιθυμείτε το λόγο, δύο λεπτά για κάθε έναν εκπρόσωπο των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Κασπάρη από το ΕΛΚ για ένα σύντομο σχόλιο ή ερώτηση που ενδεχομένως θέλετε να θέσετε στον Επίτροπο. Ähm, Αξιότιμε Πρόεδρε, Έβαλα πιο αργά να δουλεύει το ρολόι, για να μην τελειώσουν γρήγορα τα δύο λεπτά. Αστείο. Χαίρομαι που ήρθε ε, πιτούτης για να μας παρουσιάσει τη νέα στρατηγική. Είναι ένα σήμα το οποίο ε, εκτιμούμε όλος ιδιαιτέρως. Ευχαριστούμε και πάλι. Η στρατηγική σας συνεχίζει τη μέχρι τούδε ισχύουσα και αν κατάλαβα καλά τη συμπληρώσατε κατά τα σημεία που ήταν σημαντικά μετά τη Λισαβόνα, νέες εξουσίες του Κοινοβουλίου και πρόσθετα θέματα ε, όπως εξωτερικές άμεσες επενδύσεις κλπ. Θα ήθελα να είχαμε επικεντρωθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια σε μια στρατηγική ε, που δεν θα έπρεπε μόνο να ισχύει επί χάρτου, αλλά να εφαρμόζεται στην πράξη. Ε, βέβαια αυτό αφορά και τους δύο προκατόχους σας οι οποίοι έθεσαν ωραίους στόχους που βρήκαν σύμφωνο και το Κοινοβούλιο αλλά η εφαρμογή έπασχε. Ε, δεν, μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί ε, κάποια συμφωνία ενισχύει μετά τις διαπραγματεύσεις των ΠΟΕ. Η διατλαντική συνεργασία δεν προχώρησε πολύ. Δεν ε, ε, σημειώσαμε επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Εσωτερικές, εξωτερικές πολιτικές δεν τις προσαρμόσαμε καλύτερα μεταξύ τους και γι' αυτό χαίρομαι πολύ που ανακοινώσατε ότι μαζί με τον αρμόδιο για την εσωτερική αγορά επίτροπο θα καταπιαστείτε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες με το θέμα. Επίσης, οι εμπορικοί μας εταίροι πώς εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Αυτό θα είναι τα επόμενα χρόνια ένα κεντρικό θέμα και χαίρομαι που αναφερθήκατε σε αυτό. Το βασικό θέμα για μένα είναι πρόκειται για εμπορική στρατηγική ή και εμπορική τακτική. Τι εννοώ. Μια στρατηγική για το εμπόριο θα πρέπει να βλέπει τον κόσμο και πώς θα είναι, όχι αύριο, αλλά μετά από 10 και 20 χρόνια. Από τη δική μου τη σκοπιά το βασικό μου ζήτημα είναι η στρατηγική που μας παρουσιάζεται, υπησέρχεται σε αυτό το ζήτημα, με αλλαγές που θα δούμε στο, στην παγκόσμια οικονομία τα επόμενα χρόνια. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον αλλαγμένο κόσμο τι ρόλο θα παίξουμε μπορούμε να χρησιμοποιούμε και στο μέλλον τις προηγούμενες εμπορικές στρατηγικές μας ή πρέπει να αντιδράσουμε με τρόπο διαφοροποιημένο. Επίσης ως εισηγητή στο Κοινοβούλιο ενδιαφέρομαι πολύ να συζητήσω με τους σκιώδη εισηγητές και ανακοινώνω ότι θα ήθελα να καλέσω τους ισχυώδεις εισηγητές στο Στρασβούργο την, επόμενη, την επόμενη εβδομάδα για μια πρώτη συνάντηση, ούτω ώστε να ε, προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια ευρεία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Και εγώ ω εισηγητή θα κάνω το πάνω, ούτω ώστε να δώσουμε μια προσήκουσα απάντηση στην πρωτοβουλία σα. Ευχαριστούμε γιατί και πάλι και προσβλέπω και εύχομαι να έχουμε στο Κοινοβούλιο μια, μια επικοδομητική και καρποφόρο συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Κάντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ. Μ' ακούτε? Σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσατε αυτό το έγγραφο. Δεν θα ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση, αλλά έχω κάποια ερωτηματικά. Ξέρετε ότι διαφωνούμε σε σχέση με την επιτυχία όχι του Global Europe. Ξέρετε ότι εμείς συμφωνούμε ότι δεν καλύφθηκαν οι προτεραιότητες που είχαν τεθεί από τους προκατόχους σας, κυρίως σε ό,τι αφορά τις επιλογές που έγιναν για τις υπηρεσίες. Ε, δηλαδή να θεωρούσαμε ότι οι υπηρεσίες ήταν προτεραιότητα για μας, όμως δεν έχουμε ακόμα αξιολογήσει τον αντίκτυπο στην απασχόληση σκοπεύετε να το πράξετε ή όχι. Η δεύτερη ερώτηση και είναι η εξή. Πώς ε, θα εντάξετε τη βιομηχανική πολιτική στον τομέα του εμπορίου. Έχετε κάποιες συγκεκριμένε ε, ιδέες, γιατί εδώ θεωρώ ότι υπάρχει σημαντική δυναμική για τη δημιουργία θέσεων εργασία. και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για μα. Τρίτο στοιχείο η ερώτηση που είναι κάτι που αφορά περισσότερο την πραγματικότητα. Αναφερθήκαμε στις διατλαντικές ε, σχέσεις ε, ποιες ε, είναι οι επιπτώσεις των πολιτικών αλλαγών ε, που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ ε, στο Βουλή των Προσώπων και τι επιπτώσεις έχουν αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Διατλαντική αγορά, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο κύριος Στάρντι από το ECR Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ. Τρία θέματα. Καταρχήν, αν ε, εννοείτε το ότι θέλετε να καταπολεμήσετε τον προστατευτισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να έχουμε νομοθεσία αντι-dumping ε, και μη δεσμολογικά εμπόδια. Αν όμως το εννοείτε, πότε προβλέπετε την αναθεώρηση των μηχανισμών εμπορικής άμυνας Δεύτερον, αναφέρεται και σωστά τις υπηρεσίες βλέπετε να υπάρχει ε, ουσιαστικά νέα δυνατότητα να εισαγάγουμε τις υπηρεσίες ε, στο γύρο της Ντόχα, γιατί περισσότεροι εδώ θεωρώ ότι ευνοούν τις πολυμερείς και όχι τις διμερείς συμφωνίες. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι πολυμερείς συμφωνίες, αλλά εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται το γύρο της Ντόχα και τέλος η αλλαγή στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, μετά τις εκλογές. Ε, έχετε συζητήσει με τους Αμερικανούς και πώς θεωρείτε ότι θα έχει επίπτωση αυτό στις μελλοντικέ εμπορικές συναλλαγές. Γιατί όποτε παραβρεθήκαμε στι συναντήσεις στο Χονγκ Κόνγκ, ε, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε φαίνεται να έχουν ηγετική θέση. Θα δούμε αλλαγές στην πολιτική του. Τώρα αισθάνεστε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω, Επίτροπε. Αναφέρεστε στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασία και σε μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσω του εμπορίου. Όμως, ε, ε, η Κομισιόν, ε, όπως ε, βάσει και του κύριου ε, του κύριου Ρέν ε, δίνει πάρα πολλά κονδύλια ε, για να σώσει τις τράπεζες και υποσκάπτει και υπονομεύει το επίπεδο ζωής πολλών ανθρώπων. Πώς αυτό συνάδει με τη δική σας δέσμευση να δημιουργήσετε περισσότερες θέσεις εργασίας όταν θα δούμε ότι θα επιδεινωθεί η ανεργία και το ίδιο και στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και πώς η δική σας δέσμευση να δημιουργήσετε θέσεις εργασίας συνάδει ε, με το ότι ε, η Κομισιόν θα ε, ουσιαστικά ευνοήσει όλα αυτά τα παράσιτα που θέλουν να ρουφήξουν το αίμα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου και όλα αυτά φυσικά επιτρέπουν την άνοδο της ενεργείας. Ε, δεν βλέπετε να υπάρχει εδώ θεμελιώδης αντίθεση σε αυτά, γιατί εκατομμύρια ε, θέσεις εργασίας μπορούν να θυσιαστούν τώρα ε, βάσει των δικαιωμάτων που δίνετε εσείς σε αυτούς τους καρχαρίες και στους κερδοσκόπους ε, στις ε, χρηματαγορές μέσω των ε, υπηρεσιών ε, που θα δημιουργηθούν. Ε, δεύτερη ερώτηση. Αναφέρεται στο έγγραφο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το αναφέρετε και εσεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν πτυχή τη εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας ρωτήσω γιατί το ο πρόεδρος Μπαρόσο πριν δύο εβδομάδες όταν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Καζακστάν, τον κύριο Νασβάγεφ, Ε, δεν αντέδρασε ε, και καλωσόρισε αυτή την δικτατορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έκανε ούτε μία κριτική για τα δρακόντια καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Καζακστάν. Ε, και είδαμε τι συνέβη σε αυτή τη χώρα Μόλι πριν δύο μήνε δηλαδή δεν υπήρξαν πολιτικά δικαιώματα, ε, καταπατήθηκαν τα εργασιακά δικαιώματα, υπήρξαν κτηνοδίε τη φυλακή ε, όλα αυτά τα θέματα, ε, όλες αυτά τα γεγονότα έλαβαν χώρα πριν από τη συνάντηση του Προεδρού Μπαρόσο με τον Προεδρό Καζακστάν και τίποτα δεν αναφέρθηκε. Ούτε μία κριτική δεν έγινε. Ε, μήπως γιατί θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πετρέλαιο και το αέριο. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, λέει ο Πρόεδρος. William Dartman από... Speroni is here. Okay. He is going to work. Grazie. Our colleague Speroni. Grazie, Presidente. Ringrazio. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Θα κάνω μια ερώτηση όχι για το κύριο θέμα της παρουσίασή σας, αλλά θέλω να αναφερθώ σε κάτι που ούτως ή άλλως επισέρχεται, γιατί ο Επιτρόπος αναφέρθηκε σε θέσεις εργασίας και θα ήθελα να αναφέρω το θέμα της μείωσης των δεσμών ε, των προϊόντων που εισαγαγούμε από το Πακιστάν ως ε, στήριξη, ως μέσο στήριξης της χώρας αυτής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Εντάξει, να συμφωνούμε με το να ε, στηρίζουμε τις χώρες που είναι σε δυσκολία, αλλά αυτό έχει και αντίκτυπο στη δική μας οικονομία στη συνέχεια, γιατί ορισμένες ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα ζημιωθούν από το μέτρο αυτό και Ίσως ε, όσα θα δοθούν στο Πακιστάν ε, θα ε, αντικατοπτριστούν εδώ ως απώλεια θέσης εργασίας στην Ευρώπη. Σκεφτείτε την βορειοανατολική Ιταλία. Εκεί έχουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις παρόμοιες με αυτές που έχουμε στο Πακιστάν οι οποίες θα θυγούν από τα μέτρα αυτά. Έτσι λοιπόν δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποιου άλλου τρόπου να βοηθήσουμε τι χώρε που έχουν πληγεί από φυσικέ καταστροφέ, χωρί να λαμβάνουμε μέτρα που θα έχουν ε, αντίκτυπο την απώλεια θέσεων εργασία στην επικράτειά μα. Ο κ. Λάιμον. Αλλά ε, θα σας δώσω μόνο ένα λεπτό γιατί αυτό είναι εξαίρεση στον κανόνα που έθεσε. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε, Επίτροπε, στις ε, ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών με τις όμορες χώρες. Αναφέρατε τη Ρωσία και αναφέρατε ότι η συμμετοχή της Ρωσίας ε, στον ΠΟΕ. Ε, η ερώτησή μου έχει να κάνει με την Ουκρανία που αναφέρεται και με τη Γεωργία. Οι συμφωνίες πλήρης, ελεύθερων, πλήρης συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ως τμήμα αυτής της συμφωνίας σύνδεσης. Η Γεωργία περιμένει, παραδείγματο χάρη, το μήνυμα ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία. Τι θα μπορούσε να περιμένει στο εγγύς μέλλον. Κύριε που έχετε το λόγο για να σχολιάσετε τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κασπάρη, έχετε δίκιο, νομίζω, ότι μπορούμε να διαφοροποιήσουμε μεταξύ στρατηγικής και τακτικής, αλλά σε τελευταία ανάλυση το θέμα αφορά την εφαρμογή. Γι' αυτό δεν διαφοροποίησα πολύ. Εφαρμογή αυτών που διαπραγματευόμαστε. Αυτό είναι η κατεξοχήν προτεραιότητα γιατί πρέπει να μας λαμβάνουν υπόψη και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όταν γράφουμε κάτι επί χάρτου θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να ανταποκριθούν στις αποφάσεις μας και να τις εφαρμόσουν. Πράγμα όχι πάντα εύκολο, αλλά οπωσδήποτε είμαστε και εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα μέσα ως Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για να τα καταφέρουμε και θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Εδώ μιλάμε για μια στρατηγική η οποία προσπαθεί να προβλέψει την κατάσταση σε όλο τον πλανήτη μετά από 5 και 10 χρόνια. Και εμείς θα πρέπει να τοποθετηθούμε εν ώψη των εξελίξεων. Γι' αυτό είπα ότι δεν πρέπει να διαφοροποιούμε πολύ μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πτυχής των πολιτικών μας, γιατί η εμπορική πολιτική πρέπει να εδράζεται στα τεκτενόμενα στην εσωτερική αγορά. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η προστιθέμενη αξία η μεγάλη της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020, όπου θα πρέπει να την εφαρμόσουμε και για μας. Αυτό δεν το κάνουμε πάντα για τη στρατηγική, με τη στρατηγική της Λισαβόνας που είναι καλή. Αν τη διαβάσετε, έχει πολύ νόημα, αλλά οφείλουμε να συμπεράνουμε ότι πολλά από αυτά που γράφουμε δεν τα εφαρμόζουμε. Εφαρμογή λοιπόν στο εσωτερικό, στο εξωτερικό είναι μέσα που μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Η σχέση μεταξύ βιομηχανικής πολιτικής και εμπορίου ε, έχει ως υπεύθυνο τον Επίτροπο Ταγιάννη, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την βιομηχανική πολιτική, όπως είπα και στην παρουσίασή μου, όπου θα εργαστεί για να εκπονήσει μέσα στο επόμενο έτος μια ανακοίνωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, στην παγκόσμια αγορά. Και επίσης είναι θέμα ε, αρμοδιοτήτων Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσαφηνίσουν τη σχετική πολιτική. Τώρα δεν πρόκειται να συζητήσω πάνω στις λεπτομέρειες αυτής της βιομηχανικής ε, πολιτικής, ε, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, αλλά έχει πολύ ε, σημαντικό σύνδεσμο με το εμπόριο. Δέστε το πρόβλημα των εξαγωγών γιατί υπήρξε πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχε σοβαρή εξωτερική, πολιτική εξαγωγών, δεν υπήρχαν σοβαρές προβλέψεις κτλ. Οπότε ποια θα είναι η επίπτωση ε, των ε, ε, μεσοπρόθεσμων ε, εκλογών για τους ε, εκπροσώπους στη Γερουσία. Έχω διαβάσει πάρα πολλά άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα που πηγαίνουν προς διάφορες κατευθύνσεις και θα επισκεφτώ τις Ηνωμένε Πολιτείε τον επόμενο μήνα. Εκεί νομίζω ότι θα αποκτήσω μια πιο συγκεκριμένη άποψη για το γενικό κλίμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει πάρα πολύ αυτό το γενικό κλίμα προσωπικά γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί δισταγμοί ε, για το θέμα του διεθνούς εμπορίου ειδικά υπάρχουν διάφορες τάσεις προστατευτικού χαρακτήρα και στα δύο μεγάλα κόμματα και στους δύο μεγάλους σχηματισμούς. Κοιτάξτε για παράδειγμα τι γίνεται ε, με, το πάρα πολύ προστατευτικό Tea Party και δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε ότι το Κογκρέσο θα αλλάξει τα πράγματα ε, σε σχέση με την ε, ανοιχτή αγορά, το διεθνές εμπόριο ε, και ότι θα κάνει μεγάλη προσπάθεια για να περατωθεί ο γύρος της Ντόχα. Νομίζω ότι αυτές οι πιέσεις αν υπάρξουν θα προέλθουν από αλλού, δηλαδή πιο συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διάφορους άλλους συμμετέχοντες του G20. Πραγματικά προσδοκώ ιδιαιτέρως να ε, δω τι θα γίνει ή τι δεν θα γίνει αν θέλετε σε αυτό το γύρο και πιστεύω ότι θα πρέπει να συγκαλέσουμε, είναι μία από τις προθέσεις μας εξάλλου, μια υπουργική συνάντηση ε, ε, σε επίπεδο G5 δηλαδή των πιο σημαντικών εταίρων για τις διαπραγματεύσεις ε, μέχρι το τέλος, ίσως όχι μέχρι το τέλος του έτους γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά στην αρχή του επόμενου έτους, ούτω ώστε να υπάρξει μια όθηση από δική μας πλευράς σε αυτές τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Κύριε Στέντι, δεν έχουμε επί του παρόντος το σχέδιο να αλλάξουμε τα συστήματα άμυνας. Τώρα, για προστασία εμπορίου. Εδώ δεν θα αναλάβουμε άμεσα δράση με την έννοια ότι δεν υπάρχει άμεση ωφελημότητα. Έχουμε ήδη τους μηχανισμούς που χρειάζομαστε. Όμως οι αποφάσεις επιτροπολογίας, και αυτό είναι σημαντικό για μας, για τις πρωτοβουλίες ε, εμπορικής άμυνας, ε, θα μας στηρίξουν, ώστε να μην είμαστε υπό την αιγίδα ενός συμβουλίου που θα αποφασίζει με ε, απλή πλειοψηφία, για παράδειγμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν θα έχουμε αυτές τις δυνατότητες, μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται με τους παρόντες μηχανισμούς και μέσα. Όταν τελειώσει ο γύρος της Ντόχα, θα δούμε τα νέα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Τώρα όμως δεν υπάρχουν σχέδια για κάτι τέτοιο, αφού δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Η Ντόχα μπορεί να ξεκλειδώσει με ένα κεφάλαιο για τις υπηρεσίες πιο συγκεκριμένο. Πράγματι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ε, μπορούμε Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στην άμα, αλλά τώρα έχει κλειδώσει η Ντόχα γιατί, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος εταίρος που μετέχει εκεί και που δεν έχει πιστεί για τη χρησιμότητα της Δόχα. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος. Αν όλοι οι βασικοί πέντε ε, πιστούν ότι έχουν νόημα όλα αυτά, εντάξει μπορούν να υπάρξουν διάφορες ιδέες για το πώς θα χρησιμεύσει καλύτερα για τον καθένα τους. Και έχουμε εκεί αντισταθμίσματα και διαπραγματεύσεις. Αλλά εδώ η διαφορά είναι ότι ένας μεγάλος εταίρος οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν πιστεί για τη χρησιμότητα της Δόχα. Πάμε να τους πείσουμε, γιατί το πιστεύουμε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε το κλίμα όχι μόνο του κεφαλαίου, αλλά και το κλίμα που επικρατεί στην κυβέρνηση και στο Καπιτόλιο. Ε, αλλιώς μπορούμε να βρούμε κανόνες και συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί σε διάφορα επίπεδα αν θέλετε. Αλλά καταρχήν πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη συμφωνία ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε. Να κάτσουμε κάτω και να διαπραγματευτούμε. Και αυτό ακόμα δεν έχει οριμάσει. Α, για το κογκρέσο τον είπα, είπα. Κύριε Χίγκινς. Με ε, πολύ αυτά που είπατε και θα μπορούσα να σας δώσω τη γνώμη μου για τη διάσωση των τραπεζών στην Ιρλανδία. Αλλά αν αυτό έχει άμεση σχέση σχετικά με την ανακοίνωσή μου για το εμπόριο δεν το ξέρω. Πριν γίνω μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχα αναλάβει διάφορες ευθύνες ως Υπουργός Εξωτερικών και ε, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης στη χώρα μου και ασχολήθηκα και με το θέμα της οικονομικής κρίσης, της χρηματοοικονομικής κρίσης. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ δύσκολο μια κυβέρνηση να αρνηθεί να σώσει τις τράπεζές της, γιατί αν δεν γίνει αυτό θα υπάρξουν ε, οικονομικά παρεπόμενα ακόμα χειρότερα από τη διάσωση. Και αν το δείτε, βέβαια αν το δείτε μέσα από το πρίσμα της διάσωσης και της υποβοήθησης του καπιταλισμού, γιατί έτσι το βλέπετε εσείς, είναι υπεραπλούστευση. Δεν μπορούμε να πούμε «Α, ε, ας τους αφήσουμε να χρεοκοπήσουν ε, τους τραπεζίτες και να δούμε τι θα γίνει» καθώς προχωράει η κρίση, όλοι ξε... φαντάζονται τι μπορεί να γίνει. Οπότε πρέπει να κάνετε μια επιλογή και η επιλογή της Ιρλανδικής κυβέρνησης αυτή ήταν. Τώρα, εσείς μπορείτε να σκεφτείτε τι εναλλακτική είχαν, αν είχαν. Και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το Καζαχστάν, έχω πάει πολλές φορές στο Καζαχστάν και το Καζαχστάν σίγουρα δεν είναι δυτικού τύπου δημοκρατία, ούτε νομίζω ότι θα γίνει τέτοιου τύπου δημοκρατία την επόμενη δεκαετία. Επίσης, ε, όμως δεν αληθεύει ότι δεν κάνουν τίποτα για αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, σε σχέση με τις θρησκευτικές πεπιθήσεις έχουν καλή προσέγγιση. Τώρα έχουν την έδρα του ΟΑΣΕ που ήταν δύσκολη απόφαση να τη λάβουμε αν θα συμφωνούσαμε να αναλάβει την έδρα του ΟΑΣΕ το Καζαχστάν. Εγώ ήμουν, υπήρξα ε, ως Υπουργός Εξωτερικών Πρόεδρος και ξέρω πώς λειτουργεί ο Τις ξέρω όλες αυτές τις συζητήσεις, αν είμαστε έτοιμοι ή όχι να βάλουμε το Καζαχστάν να αναλάβει ενεργά την Προεδρία. Αλλά σε τελευταία ανάλυση καλά κάναμε, γιατί κάνουν καλή δουλειά και αν θέλουμε να αναπτυχθεί ο ΑΣΕ και στο μέλλον θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Δεν μπορεί να έχουμε δηλαδή ο ΑΣΕ ο οποίος θα προεδρεύεται πάντοτε από ευρωπαϊκές χώρες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα γιατί τότε θα αποδυναμωθεί ο οργανισμός. Οπότε αυτή και σίγουρα γίνεται δουλειά προοδεύουν. Σε άλλους τομείς επιτελούν περισσότερη πρόοδο, αλλού όχι. Λέτε ότι έχει το αέριο. Ε, υπάρχει πολύ αέριο και σε άλλες χώρες. Δηλαδή δεν είναι ότι χωρίς το Καζαχστάν δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν, ούτε οι εισαγωγές μας από εκεί είναι τόσο μεγάλες. Καλύτερα είναι να αυξήσουμε τις εισαγωγές γιατί δεν θα πρέπει να εξαρτώμεθα από μια χώρα για ε, εισαγωγές αερίου. Τα έχουμε δει αυτά. Μέσα περιπτώσει όλα αυτά τα θέματα ε, δημιουργούν μια πιο σύνθετη εικόνα από αυτή που μας παρουσιάσατε εσείς. Βέβαια το πλεονέκτημα είναι ότι τα είπατε απλά. Και μου άρεσαν οι ερωτήσεις για το Πακιστάν, κύριε Σπυρώνε. Αυτό το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Πρέπει να φύγω κιόλα σε κάνα δυο λεπτά, γιατί στις 12 έχω μια παρουσίαση. Αυτό που προτείναμε είναι ένα συμβιβασμός η καλύτερη απόδειξη ότι είναι συμβιβασμός είναι ότι κανεί δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχή, ούτε το Πακιστάν ούτε οι Ευρωπαίοι. Και τώρα ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσουν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση, εκλήθη, θα κάνουμε μια μετριοπαθή αλλά και ουσιαστική πρόταση. Αυτό ζητήθηκε. Τώρα η επίπτωση στην ευρωπαϊκή οικονομία και τις θέσεις εργασίας έχει ε, πολύ ε, υπερτονιστεί, καθ' δηλαδή, γιατί είναι μόνο γύρω στα 15 εκατομμύρια πρόσθετες αγωγές. Και βέβαια, αν υπάρχει ε, επίπτωση σε 100.000 θέσεις εργασίας, αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Ε, για την Ρωσία και την κυρία Αντρικιένα. Έχουμε κάποια προβλήματα ακόμα με τη Ρωσία, αλλά νομίζω ότι με την προσχώρηση στο ΠΟΕ θα βελτιωθούν τα πράγματα. Θα είναι καλό που θα είναι στο ΠΟΕ, γιατί είχαμε στην κρίση πολλές προστατευτικές κινήσεις, ακριβώς επειδή δεν ε, ε, είχαν ανάγκη να σέβονται τους κανόνες του ΠΟΕ. Βέβαια έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τη Ρωσία ακόμα σχετικά με τους εξαγωγικούς δασμούς και για την Γεωργία και την Ουκρανία. Πήγα στην Ουκρανία πριν από 10 μέρες. Εκεί ήμουνα. Θέλουμε να καταλήξουμε και με τη Γεωργία σε μια συμφωνία. Ε, επετέλεσαν πρόοδο τελευταία γιατί πέτυχαν τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης που είχαμε θέσει. Πολλά μέλουν ακόμα να γίνουν και επίσης υπάρχουν και περιορισμοί ικανοτήτων από την πλευρά τους. Είναι περιορισμένες οι ικανότητές τους, οπότε δεν πρέπει μόνο να διαπραγματευόμαστε για τον εαυτό μας, αλλά θα πρέπει να δίνουμε και τεχνική υποστήριξη σε εκείνους για να έχουμε μια συνεκτική Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών ε, και με την Ουκρανία. Ε, η Ουκρανία πιέζει και συζητήσαμε αρκετέ ώρες με τον Πρωθυπουργό Αζάροφ όταν πήγα στο Κίεβο. Οπότε δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Εμείς θέλουμε συμφωνίε μαζί τους, θέλουμε να επιδείξουμε ευελιξία, αλλά και εκείνοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά που του αναλογεί. Ε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανακοίνωση και Βεβαίως ε, ήταν πάρα πολύ ε, ενδιαφέροντα όσα μας είπατε, όπως φάνηκε και από, το από την εκτενέστατη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ. Ας προχωρήσουμε χωρίς χρονοτριβή στο επόμενο ζήτημα. Item number 9. Σημείο 9. Εφαρμογή ορισμένων κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τη χάνουν δημόσια στήριξη. Σας παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την προσοχή σα όσοι εγκαταλείπουν την αίθουσα. Παρακαλώ να το κάνετε ταχύτερο. And please don't hold, do not hold conversations in the room. Σας παρακαλώ μη συζητάτε στην αίθουσα. So, item number nine, application. Σημείο 9, λοιπόν, εφαρμογή κατευθυντηριών γραμμών στον τομέα εξωγικών περιστάσεων που διχανούν δημόσια στήριξη. Θα εξετάσουμε την ε, έκθεση του κυρίου Ζαντό για το πώς θα συμπεριλάβουμε αυτούς τους ε, χρηματοδοτικούς κανόνες ε, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είμαστε η Καθελήν Επιτροπή. Εισηγητής είναι ο κύριος Γιάννη Ζαντό από τους Πρασίνους. Έχετε το λόγο, Γιάννη. Σας παρακαλώ, θα ήθελα να είστε προσεκτικοί. Και you can... Merci, Monsieur le Président. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε φτάνουμε στο πέρας ε, της ε, διαδικασίας εξέτασης από το Κοινοβούλιο. Αυτού του νομοθετικού ψηφίσματος το επιθυμήσατε. και έτσι οι νέες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και αυτής της Επιτροπής ε, τοποθετούνται σε σχέση με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές του ΣΟΝΤΕΟ έχουμε μια συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών και θα ήθελα να υπενθυμίσω ορισμένα σημεία πάνω σε αυτή την εισήγηση και να διευκρινίσω διάφορες προθέσεις από δική μου πλευράς. Καταρχήν έχουμε μια σειρά από τροπολογίες οι οποίες προτείνονται σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αφορά αποκλειστικά ε, τίματα επιπρόσθετα σε θέματα reporting. Τώρα, το θέμα δεν είναι να δημιουργήσουμε φόρτο διοικητικό για τα κράτη-μέλη ε, και για, τα, για τους οργανισμούς εξαγωγών. Επίσης δεν θέλουμε να επινοήσουμε νέα κριτήρια που θα πλαισιώνουν αυτές, ε, αυτά τα γραφεία ε, αλλά πιστεύουμε ότι επειδή υπήρξε η χρηματοοικονομική κρίση, επειδή υπάρχει μια ανησυχία από πλευράς Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα ε, οικονομικά των κρατών και τις, ε, ε, τα προβλήματα όλων των χωρών μελών της Ευρώπης. Πιστεύουμε λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες αυτές τις δραστηριότητες της του οργανισμού ε, πιστώσεων ε, πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του οργανισμού αυτού. Θα ήθελα να τονίσω τα εξής. Ε, στον υπολογισμό των κινδύνων ε, ορισμένων σχεδίων δεν υπάρχουν μόνο οι διαστάσεις του εμπορικού ή του πολιτικού κινδύνου. Ξέρουμε ότι πάνω σε μια σειρά σχεδίων, κάτι το οποίο επισέρχεται στη συζήτηση για τα σχετικά σχέδια ε, όταν υποβάλλονται προς έγκριση, υπάρχουν και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και οι κοινωνικοί κίνδυνοι. Και ακριβώς για να υπάρχει σωστή χρηστή διαχείριση όλων αυτών των οργανισμών θέλουμε να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, γίνεται ο υπολογισμός των επιδοτήσεων και επίσης τι ε, πώς γίνονται οι εγκρίσεις, ε, με βάση ποιον υπολογισμό του κινδύνου. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό γιατί ευνοεί την διαφάνεια. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια. Υπάρχει επίσης μια δεύτερη συστάδα τροπολογιών. Προτείνουμε μέσα από αυτές τις τροπολογίες να συνεργαστούν αυτοί οι οργανισμοί εξαγωγών με και να προσαρμοστούν προς τους στόχους της συνθήκης της Λισαβόνας, όλους τους στόχους και τις προδιαγραφές για το περιβάλλον, είτε είναι για το περιβάλλον, είτε είναι κοινωνικοί στόχοι, είτε είναι... Ε, στόχοι γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους συμμετέχουν και οι χώρες του G20 για το περιβάλλον και για διάφορες συνέργειες ε, πιστεύουμε ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα προβλήματα, νέα κριτήρια, νέες ε, οθήσεις. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι ενεργά αυτά τα κριτήρια μέσα στους υπάρχοντες ε, οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων, ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, ούτως ώστε και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή και το Συμβούλιο να μπορούν να έχουν μια χρηστή διαχείριση ε, των ε, ε, δημοσιονομικών πόρων και να έχουν μια συνεκτικότητα οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται ένα θέμα το οποίο ίσως να το παρατηρήσατε στην εισήγηση που προτείνουμε ότι υπάρχει μία πράξη της αντιπροσωπείας εξ ονόματος της Επιτροπής. Είπα από την αρχή ότι ήμουν υπέρ, ιδιαίτερα υπέρ, στο να μην είμαστε υποχρεωμένοι μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς να επιτελέσουμε όλη την εργασία της επικύρωσης των προτάσεων της Επιτροπής ε, και να ε, ε, κάνουμε εμείς την ε, εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του ε, ΟΣΑ. Πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει περισσότερη διαφάνεια σε σχέση με, τους, ε, με τις εξαγωγικές πιστώσεις και τους σχετικούς οργανισμούς. Εάν υπάρξει αυτή η διαφάνεια τότε θα έχουμε μεγάλη διευκόλυνση και εμείς για τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. Έχουμε στην περίπτωση μας ε, την εισαγωγή των κατευθυντηρίων γραμμών του 2005. Ε, οπότε οι κατευθυντήριες γραμμές του 2011 ε, επί του παρόντος είναι στα, διαπραγματεύσιμες και υπάρχει διαπραγμάτευση και εκεί επισέρχονται και οι δείκτες για το περιβάλλον. Τι θέλουμε εμείς με την διαφάνεια. Ε, με τη διαφάνεια διευκολύνεται η μεταφορά των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΣΑ ε, ούτως ώστε να υπάρχει μια καλύτερη ε, ε, επιτέλεση των καθηκόντων μας σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές του 2011. Τώρα θέλω να σας πω δύο λόγια και για την Κίνα κύριε Πρόεδρε. Τι κάνουμε ε, ε, με την ε, διαφάνεια τη μεγαλύτερη την οποία επιβάλλουμε στις, στους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων σε σχέση με την Κίνα μήπως κάνουμε κακό στον εαυτό μας όχι πιστεύω ότι πρέπει μέσα στα υπάρχοντα σημερινά πλαίσια να καταλάβουμε βεβαίως ότι η Κίνα είναι πολύ επιθετική φαίνεται πολύ επιθετική μέσα από την προαγωγή των νομισμάτων της ή μέσα από τον τρόπο που προωθεί τις εξαγωγές της ναι αλλά πρέπει πιστεύουμε να οθήσουμε την Κίνα να υιοθετήσει τα κριτήρια τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τον ΩΣΑ και μόνον έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια νέα όθηση εξελικτική σε αυτόν τον νέο τομέα ε, που θα είναι ωφέλιμη για μας. Θα ήθελα περατώντας κύριε Πρόεδρε να ζητήσω μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων, κάτι που δεν υπάρχει στα κράτη-μέλη, καλύτερη διαχείριση των ε, ευρωπαϊκών ε, πόρων, δημοσιονομικών πόρων ε, και επίσης για τα θέματα τα κοινωνικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος θα πρέπει να εγγραφούν στους στόχους των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων. Ε, αυτά ζητάμε και τίποτα παραπάνω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα ε, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής κύριο Βέρνεν Σόλτς ειδικά για τις ε, τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής. Καταρχήν, να τονίσω ότι συμφωνεί απόλυτα η Κομισιόν ότι χρειάζεται σωστή επιτήρηση αυτής της πολιτικής, ενώ απ' την άλλη πρέπει να αξιοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο τους υφιστάμενους μηχανισμούς χωρίς επικαλύψεις και πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τους εμπλεκομένους. Για μας, οπωσδήποτε, το σημαντικότερο ζήτημα είναι η διαφάνεια και η υποβολή εκθέσεων. Η Κομισιόν συμμερίζεται απόλυτα την ιδέα ότι πρέπει να επεξεργαστούμε ένα σωστό μηχανισμό για κάτι τέτοιο. Έχουμε κάπως την εντύπωση ότι οι τωρινές τροπολογίες μπορεί να πρέπει να δουλευτούν κι άλλο για να λύσουμε τεχνικά και πρακτικά θέματα. Σας θυμίζω ότι αυτή δεν είναι μια πολιτική στην οποία η Κομισιόν έχει ρόλο ε, πρακτικής εφαρμογής ε, στον Ευρωπαϊκό δεν είναι ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, είναι η εθνική προϋπολογισμοί των κρατών μελών και είναι δύσκολο να υποβάλουμε εκθέσεις εμείς για την λειτουργική επιχειρησιακή πλευρά του θέματος. Πρέπει να προέλθει από τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο. Από την άλλη, ευχαρίστως να υποβάλλουμε σε τακτά διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τους κανόνες σε όλους τους συναφείς τομείς όπως διαπραγματεύσεις, ΠΟΕ, το θέμα κρατικών ενισχύσεων που αφορούν επίσης τις εξαγωγικές πιστώσεις και την και αρμοδιότητα της Κομισιόν. Όπως είπα, βλέπουμε ανάγκη να λάβουμε υπόψη μας και τα κράτη-μέλη από κοινού πρέπει να ξαναδούμε το θέμα, ώστε να το δούμε στο σωστό πλαίσιο. Δεύτερον, για την έκδοση των για το θέμα των προτύπων, θυμίζω ότι ο ΩΣΑ έχει μια συγκεκριμένη δομή. Από τη μια υπάρχει ο διακανονισμός και από την άλλη πλευρά οι συστάσεις πολιτικής του ΩΣΑ που αφορούν τα περισσότερα θέματα πολιτικής που αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε παντελώς ε, αυτούς τους μηχανισμούς όπως διαφοροποιούνται και πρέπει να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να μεταφράσουμε τις επιθυμίες μας και για τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε αυτό το επίπεδο. Να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Οι κοινέ προσεγγίσεις που είναι τα πιο σημαντικά μέσα που έχουμε σε αυτόν τον τομέα. Ήδη τώρα περιέχουν μια διάταξη που μας επιτρέπει να έχουμε κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης έναντι ευρωπαϊκών προτύπων, σαφέστατα, Οπότε αν στη ε, συνεχιζόμενη αναθεώρηση του μέσου επιμείνουμε να διατηρηθεί η διάταξη αυτή, αυτό θα καλύψει πολλές από τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν. Επίσης σε αυτό το μέσον θα υπάρχει και μια προσθήκη ε, ε, ειδικών πολιτικών διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οπότε και πάλι το μέσον αυτό πιθανό να εξελιχθεί προς μια κατεύθυνση που θα σας καλύπτει σε επίπεδο πολιτικής. Τέλος, ακόμα κι αν αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα, εμείς θα επαναλάβουμε με στεναρότητα την ανάγκη να εξεταστεί η εναλλακτική, να υπάρχει στο μέλλον το μέσον των κατεξουσιοδότηση πράξεων για την τεχνική μεταβίβαση κανόνων και μεταφορά τους. Η κατεξουσιοδότηση πράξη δεν σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, ε, παραχωρήσουν πολιτικές εξουσίες. Είναι μια εντολή για την Κομισιόν να κάνει τεχνική ενημέρωση και παράλληλα και τα δύο θεσμικά όργανα να πάσα στιγμή μπορούν να ανακαλέσουν αυτή την κατεξουσιοδότηση πράξη χωρίς καμία δικαιολογία. Και Αυτό που θα κάνει η Κομισιόν και θα μεταφέρει σε ευρωπαϊκό δίκαιο μπορεί να ανατραπεί μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Οπότε υπάρχουν διασφαλίσεις, πολλές διασφαλίσεις, ότι δεν δημιουργείται καμία ανισορροπία εδώ μεταξύ των σχέσεων των θεσμικών οργάνων. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, κύριε Γκάσπερη, να είστε όσο γίνεται πιο σύντομος παρακαλώ. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά του εισηγητή που εντατικά αντιπαρατέθηκε με το θέμα. Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούμε όλοι ότι το θέμα είναι σύνθετότατο. Νομίζω ότι σε όλο αυτό το θέμα των εξαγωγικών πιστώσεων χρειάζεται διαφάνεια, είναι σαφές, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες έμαθα ότι στα πλαίσια του ΟΣΑ και του ΠΟΕ ήδη γίνονται πολλά για τη διαφάνεια, ιδιαίτερα στις κατευθυντήριες γραμμές που θέλουμε να μεταφέρουμε στο ευρωπαϊκό μας δίκαιο. Ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολλές διαδικασίες και πληροφοριών και ανταλλαγές πληροφοριών που μπαίνουν μέχρι και σε εξειδικευμένες περιπτώσεις και υποθέσεις. Μέσω του ΩΣΑ σήμερα περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, κοινωνικοί κίνδυνοι εξετάζονται, λαμβάνονται υπόψη ε, μέσα από έρευνες του ΟΣΑ προσανατολίζονται προς τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Τράπεζας, εν μέρη και του International Finance Corporation και στους κόλπους του ΩΣΑ. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό που με απασχολεί πολύ περισσότερο είναι το εξής θα έπρεπε να στοχεύσουμε την, την, την αναβάθμιση της, ευρω, της διαφάνειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως λέει ο συγητής, ή θα πρέπει να στοχεύσουμε αφενός οι εταίροι του οσα επιτέλους κάποια στιγμή να τηρήσουν τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τηρούν, γιατί εκεί υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στον ΩΣΑ. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι, και δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συζήτηση από αυτού, ποια είναι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα ε, των ε, χωρών και των ε, οικονομικών χώρων γιατί πολλές φορές ο ανταγωνισμός είναι σε βάρος των επιχειρήσεών μας. Βλέπε Κίνα που είναι τόσο επιθετική και βίαιη στο άνοιγμα νέων αγορών ενώ εμείς δεν έχουμε την πρόσβαση γιατί λειτουργούμε με βάση κάποιες βασικές αξίες και πεπιθήσεις. Μην με παρεξηγήσετε. Δεν θέλω να αποδυναμώσω τις, κατευθυντήριε κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ. Αντίθελα, αντίθετα θα ήθελα να ισχύουν παγκοσμίω. Αλλά θα ήταν λάθος επίσης ως Ευρωπαϊκή Ένωση κινούμεθα μονόπλευρα και κάναμε αυστηρότερους τους κανόνες μας ε, και σε περίπτωση αμφιβολιών θα γίνονται τα έργα, θα συνεχίσουν να γίνονται, αλλά θα χρηματοδοτούνται από άλλους, από ανθρώπους που δεν ε, τους ενδιαφέρει η διακυβέρνηση, δεν τους ενδιαφέρουν οι κοινωνικές αξίες, η η ε, βιωσιμότητα, αλλά τους ε, ενδιαφέρει να επιτύχουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη παραγωνίζοντας εμάς από τις αγορές. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων λοιπόν αν τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην Ολομέλεια αξιοποιούσαμε το διάστημα αυτό που μας δίνεται για να συζητήσουμε πώς μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να πείσουμε τους εταίρους των ΩΣΑ να τηρούν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν και πώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνουμε το πάνω τόσο ώστε περισσότερες χώρες στον κόσμο θα τηρούν αυτές οι παρόμοιες υποχρεώσεις πριν πάμε στο δεύτερο βήμα για να βελτιώσουμε το σύστημα που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό είναι λοιπόν να κάνουμε μια μετατόπιση του πρίσματος της επόμενης εβδομάδα και να κάνουμε αυτά που είπα. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα τρία άτομα που ζητούν το λόγο. Θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε στο δυνατόν πιο σύντομοι, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ε, θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος ε, του συναδέλφου που δεν είναι εδώ σήμερα συμφωνεί με τη φιλοσοφία της εργασίας του κυρίου Σαντό. Είναι σημαντική δουλειά. Συμφωνούμε και με τις περισσότερες ε, τροπολογίες. Πράγματι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια για τον τομέα αυτό και για τις επιδόσεις ε, των οργανισμών εξαγωγικών ε, πιστώσεων. Μάλιστα προβλέπεται και ένα οργανισμό υποβολής εκθέσεων και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τους όρους υπό τον οποίο εργάζονται αυτοί οι οργανισμοί και ποια μεθοδολογία χρησιμοποιούν. Και στα πεντέτη θα έχουμε και μια αξιολογία στο τομέα. Ίσως θα έπρεπε να προσθέσουμε μία αναφορά και στην εταιρική ευθύνη ε, των επιχειρήσεων, ε, στην κοινωνική ευθύνη των εταιριών. Θα έπρεπε να αναφερθούμε και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, οι οποίες δεν θα έπρεπε να ποινικοποιηθούν από αυτό το διακανονισμό και μάλιστα δεν θα έπρεπε να ποινικοποιηθούν έναντι των άλλων αναδυόμενων χωρών όπως ε, η Βραζιλία ή η Κίνα και θα πρέπει όλοι, όλοι να έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε και τη Συμφωνία ΩΣΑ και σε άλλες χώρες αυτά για να εργαστεί ο κύριος Ζαντό επί του θέματος αυτά. Ευχαριστώ. William Dartmouth. Ναι. Πρέπει να συγχαρώ τον κύριο Ζατό, ο οποίος ε, ξεκαθάρισε ότι εμπίπτουν οι, οι τροπολογίες του σε πολύ σαφείς κατηγορίες. Το πρώτο σύνολο τροπολογιών αναφέρονται στην ε, συνοχιζόμενο έλεγχο και στη διαφάνεια και είμαστε υπέρ και ελπίζω ο κύριος ε, Ζαντό να παρουσιάσει και την τροπολογία του στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είμαστε επέρ αυτού. Και οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ ε, θεωρώ ότι θα ψηφίσουν αυτή την, ε, αυτό το σύνολο τροπολογιών. Όμω υπάρχει και ένα άλλο σύνολο τροπολογιών που αναφέρεται στην πολιτική, που σχετίζεται με την πολιτική μα ατζέντα. Το είπα αυτό στο παρελθόν, αλλά θα το ξαναπώ. Κάποιο ε, που είναι τώρα εκλεγμένο πολιτικό δεν ε, θα έχει παρά ε, τον ε, απόλυτο θαυμασμό για την επαγγελματική δουλειά του κ. Ζαντόλα. Για κάποιον που είναι δημοκράτης, εγώ μπορώ να σας πω, δεν είμαι απόλυτα υπέρ, γιατί το Πράσινο Κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε το 9%. ενώ το 91% των ψηφοφόρων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ψήφισε για τους Πρασίνους δεν γνωρίζω τις στατιστικές ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά μπορώ να σας πω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μάλλον έχουμε 5% του συνολικού του πληθυσμού που ψηφίζει πράσινους. Τώρα τι κάνει ο κύριος ε, ε, Ζαντό σε μεγάλο επίπεδο, δηλαδή χρησιμοποιεί την έκθεση αυτή σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, ε, μπορείτε να συντομεύσετε, γιατί ήδη έχουμε περάσει στο χρόνο που θα πρέπει να αφιερώσουμε για το επόμενο θέμα, θα πρέπει να το δούμε πριν το διάλειμμα. Κοιτάξτε, ουσιαστικά χρησιμοποιεί ε, την υποστήριξη μας για να επιβάλλει μια πολιτική στρατηγική μειοψηφία. Δηλαδή αυτό το τμήμα των τροπολογιών δυστυχώς δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε, αλλά όπως πάντα θαυμάζω τον κύριο Ζαντού. Μάλιστα. <laughs> Ακούσαμε λοιπόν τις παρεμβάσεις σας. Σας παρακαλώ αυτή τη φορά να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομος, κύριε Χίγκινς. Ναι, θέλω να συμβουλεύσω τον κύριο Ζαντό είναι πολύ προσεκτικός Θεωρώ ότι το όλο θέμα των εξαγωγικών πιστώσεων ε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχείται σήμερα από αυτούς ε, που υπερασπίζουν τις ε, καπιταλιστικές αγορές, δηλαδή να μην υπάρχει κανένας κριτικός παρεμβατισμός, θέλουν να συμμετέχουν και στις δημόσιες συμβάσεις, να ιδιωτικοποιήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και οτιδήποτε άλλο μπορούν να αδράξουν. Αλλά Κάποιες από τις μεγαλύτερες συμφωνίες, από τις μεγαλύτερες εταιρείες ε, ε, βλέπουμε ότι γίνονται και με τη συμμετοχή του κράτους ε, και έχουμε και συμμετοχή των φορολογουμένων. Αυτό είναι μία αντίφαση και συνήθως σιωπούν από αυτόν οι σχολιαστές της δεξιάς. Όμως ε, απλώς προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει παρέμβαση του κράτους. Τώρα, εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Τσεντό ότι αφού συμμετέχει και το κράτος σε αυτές τις δραστηριότητε ε, και έχουμε χρήματα των φορολογουμένων που χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να έχουμε και στόχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να έχουμε και στόχους για τη βέλτιστα περιβαλλοντικά πρότυπα. Και αναφέρεται ε, το έγγραφο του κυρίου Ζαντό σε project που υποστηρίθηκαν στην περίπτωση του φράγματος ε, στην Τουρκία. Αρχικά υποστηρίχθηκαν ε, από τους οργανισμούς εξαγωγικών ε, πιστώσεων που, ε, ήταν, ε, που είναι ουσιαστικά αντίθετη στην χρήση των βελτιστών περιβαλλοντικών πρακτικών. Το γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων στη Βρετανία ε, αλλά και στην Ευρώπη θέλουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβονται και να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω και να προωθούν τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές. Και επομένως όταν ο κύριος Ζαντό αλλά και εγώ και άλλοι εδώ επιθυμούμε να συμπεριληφθούν σε τέτοιους διακονονισμούς απαιτήσει ότι θα γίνονται αυτά τα πράγματα, τελικά εδώ εκφράζουμε την άποψη της πλειοψηφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό, Πρόεδρε, αφορά κυρίω ορισμένα μεγάλα project εξωτερικά, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που αφορούν ε, το αέριο, το πετρέλαιο και αυτά τα project μπορεί να έχουν πολύ συχνά πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στους τοπικούς πληθυσμούς και πρέπει να επιμένουμε ε, σε αυτά τα ζητήματα, κυρίως όταν χρησιμοποιούμε τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογμένου. Κύριε Ζαντού, τα τελευταία σχόλια παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ και για τα κοπλιμέντα που μου απευθύνατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η εργασία σε αυτό το κοινοβούλιο ε, δεν ε, έχει να κάνει με ε, τη βαρύτητα των ψήφων που λαμβάνουμε στις χώρες μας. Ε, γιατί εδώ είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσπαθούμε να ασχοληθούμε με ευρωπαϊκά ζητήματα. Εδώ αναφερόμαστε σε πρότυπα που υπάρχουν και σε κανόνες που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, απαντούμε ε, εν μέρη στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Η ιδέα είναι να μάθουμε ποιο, πώς γίνεται ο υπολογισμός του κινδύνου, πώς γίνεται ο υπολογισμός ε, του ασφαλίστρου και αν λαμβάνονται υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια που εμπίπτουν σήμερα στην ανάλυση του κινδύνου. Δηλαδή δεν μιλάμε ακριβώς για κοινέ ε, ε, προσεγγίσεις, μιλάμε για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι χώρες αυτές. Και όταν μιλάμε για τον ε, ΟΣΑ, ε, οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων στον ΙΠΑ υποβαλούν εκθέσεις στο Κογκρέσο ε, και στον ΟΣΑ. Και έτσι ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει και μεγαλύτερη σοβαρότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κάτι ακόμη για το θέμα της Κίνας. Αυτό ξεπερνά το συγκεκριμένο φάκελο. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα δεν ε, κατορθώνουμε να έχουμε εύρωστες ε, εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. Δεν θα το κατορθώσουμε αν στην ευρωπαϊκή πολιτική δεν ε, εφαρμόσουμε τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και τους περιβαλλοντικούς κανόνες ο πρόεδρος της Κίνας και τη Γαλλία ε, αυτές τις ημέρες. Ε, ο τρόπος που θέλουμε να παραγνωρίσουμε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ε, δημοκρατίας στην Κίνα ε, οδηγεί στο να έχουμε άνισες ανταλλαγές. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να θέσουμε και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά και δημοκρατικά ζητήματα με την Κίνα, γιατί αν δεν το πράξουμε πάντα θα χάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζαντό. Προθεσμία για τις ε, τροπολογίες 12 του μηνός. Έχουμε 18 λεπτά, 20 λεπτά το πολύ. Και πρέπει να δούμε τα θέματα 13 και 14, συμφωνίες για το εμπόριο για τις μπανάνες δεύτερη φορά ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Και θα επανέλθουμε όταν θα συζητήσουμε την έκθεση δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για αυτούς τους δύο φακέλους. Η συγγήτρια και για τα δύο αυτά θέματα είναι η Φραντσέσκα Μπαλτσάνη δεν ε, μπορεί να είναι εδώ σήμερα γιατί ε, γέννησε. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητηριά μου στη μητέρα και στο παιδί και θα ακούσουμε τον αντικαταστάτη της κυρίας Μπαλτσάνη. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μου ζήτησε λοιπόν να μιλήσω η Φραντσέσκα πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο συζητείται εδώ και πολύ καιρό. Όλοι χάρηκαν πάρα πολύ για το επίτεμα του ΠΟΕ. Δεν ακούγεται καλά ο μιλητής. Όλοι λοιπόν έλεγα ότι χάρηκαν με την συμφωνία του ΠΟΕ για, τις, ε, ε, για το εμπόριο μπανάνας ήταν ε, ένα θέμα σύνθετο τεχνικά και πολύ σημαντικό εμπορικά. Ε, και υπήρχε μια διαμάχη σημαντική έτσι που μπόρεσε να την επιλύσει σωστά ο ΠΟΕ. Ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη για αυτή τη συμφωνία. Δεν είχαμε τέτοια σύμφωνη γνώμη από πλευράς Κοινοβουλίου, γιατί το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δώσει σύμφωνη γνώμη αν δεν έχει σαφείς ε, ε, δεσμεύσεις και όχι μόνο σαφείς, αλλά πολύ συγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είπαμε λοιπόν ότι χρειάζεται για τις χώρες παραγωγούς μπανάνας μια νέα συζήτηση, καθώς και για τις υπερπεριφερειακές ε, περιφέρειες. Ε, θέλουμε να υπάρξουν μέτρα συνοδευτικά για το εμπόριο μπανάνας και 18 μήνες πριν να εκπνεύσει το πρόγραμμα θα πρέπει να κατατεθεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα στο Κοινοβούλιο με τα ε, σχετικά μέτρα. Ε, δεν μπορούμε σήμερα να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία για τις χώρες ΑΚΕ. Ε, σήμερα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει μια στήριξη των παραγωγών η οποία δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί όμως από ε, ποσά που προέρχονται από αναπτυξιακά προγράμματα και επίσης οι δασμοί για τις μπανάνες θα πρέπει να, είναι, να προέρχονται από χώρες οι οποίες χάνουν μερίδια από τις εξαγωγές τους. Ε, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι δείκτες τους οποίους ε, βρήκαμε ούτως ώστε να τοποθετήσουμε σωστά το εμπόριο της μπανάνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα σημεία ε, είναι και δεσμεύσεις που ζητούμε σχετικά με τις προτεραιότητές μας. Εάν δεν έχουμε αυτές τις δεσμεύσεις δεν θα μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε και να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε ορισμένους εκπροσώπους εδώ από ε, συνδέσμους ε, ευρωπαϊκών ε, παραγωγών μπανάνας ο κύριος Ζεραρμπαλή, ο κύριος Κόνογκαν, ο κύριος Φρανσίσκο Ροντρίγκε. Είναι, ας ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε αυτό το θέμα. Ποιος θα μιλήσει από την Επιτροπή. Νόρις λέγομαι, εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με τον πρέσβη Έκον Κούτς, και για το θέμα της μπανάνας και τα κάποια συνοδευτικά μέτρα ε, κατά της διάβρωσης. Δεν θα παρουσιάσω την σημασία αυτής της συμφωνίας, ήδη τα ακούσαμε. Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε και παρουσίαση από τη γραμματεία του ΠΟΕ και κάποιον που συνεργάζεται στενά με τη Γενική Διεύθυνση και που υπογράμμισε με ωραιότερο και γλαφυρότερο τρόπο από ό,τι θα μπορούσα εγώ ποτέ πόσο σημαντική είναι η συμφωνία αυτή και πόσο σημαντικό είναι να συναυθεί το ταχύτερο δυνατόν. Κύριε Πρόεδρε, αυτή παραμένει η θέση μας και στηρίζουμε την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο που συμφωνεί επίσης. Το Συμβούλιο ομόφωνα ψήφισε υπέρ και πρέπει να το προχωρήσουμε το θέμα το ταχύτερο δυνατόν. Τώρα, πιο συγκεκριμένα να αναφερθώ στα θέματα που παρουσιάσετε σε ό,τι αφορά τη μελέτη επιπτώσεων ή αντίκτυπου κύριε Πρόεδρε βεβαίως και το είδαμε το θέμα κατά το παρελθόν για τους δικούς μας τους παραγωγούς ε, έγινε κάτι τέτοιο στα πλαίσια μάλιστα του μεταρρυθμιστικού πακέτου που μπόρεσε να διασφαλίσει ότι θα υπήρχαν κονδύλια για να συνεχιστεί η παραγωγή στον τομέα. 278 εκατομμύρια ευρώ έχουμε γράψει στον προϋπολογισμό γι' αυτό. Και όπως σας είπα, Έγιναν συζητήσεις με τους ενδιαφερομένους και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, αλλά και με βάση μια μελέτη επιπτώσεων η οποία εξέτασε πολύ προσεκτικά μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης του εμπορίου μετά από τη Συμφωνία για την Μπανάνα. Τότε δεν είχαμε όλες τις παραμέτρους υπόψη μας, αλλά μπορέσαμε να στηρίξουμε τις παραμέτρους της μελέτης επιπτώσεων ουσιαστικά ε, σε αυτά που απεδείχθη ότι ήταν και τα τελικά οριστικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις περικοπές των δασμών. Οπότε είμαστε, πέσαμε πολύ κοντά και θα έλεγα ότι είμαστε, υπήρξαμε και πιο απεσιόδοξοι. Οπότε νιώθουμε πολύ καλά μετά από τη μελέτη επιπτώσεων. Τώρα, για τις ΑΚΕ Το είδαμε το θέμα, κάναμε και διαμακρών συζητήσεις με τους εταίρους μας από τις χώρες ΑΚΕ, συμμετείχαν πλήρως και νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό είναι ένα πακέτο που τους ενδιέφερε και εκείνους σε ό,τι αφορά δηλαδή το θέμα των διαβρώσεων των προτιμήσεων που είναι πολύ σημαντικό θέμα για τις ΑΚΕ στον ΟΜΠΟΕ απλούστατα διότι με την απελευθέρωση του εμπορίου σιγά σιγά διαβρώνονται οι προτιμήσεις που έχουν οι χώρες ΑΚΕ και είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα μέσα, και να το λύσουμε μέσα από διάφορα άλλα μέτρα και αυτό μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το πακέτο για τη διάβρωση των προτιμήσεων. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο και βοήθησε θα έλεγα τις χώρες ΑΚΕ να ενταχθούν στο πακέτο και να συμφωνήσουν και όλοι συμφώνησαν πάνω στη βάση ενός ε, πακέτου με τροπικά προϊόντα, διάβρωση των προτιμήσεων και τις μπανάνες. Οπότε νιώθουμε άνετα ότι τα συμφέροντα των ΑΚΕ ελήφθησαν απόλυτα υπόψη ε, εδώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Αντρικένε από το ΕΛΚ. Μας λείπει χρόνος, τελειώνει ο χρόνος. Παρακαλώ, σύντομα, δύο λεπτά να προτείνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ η συγγήτρια Φραντσέσκα Μπαλσάνη δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Ε, για καλό σκοπό όμω, τη ευχόμεθα το καλύτερο. Τώρα συζητάμε δύο εκθέσει. Η μία αφορά τη Συμφωνία για την Πανάνα του ΠΟΕ και το άλλο είναι οι επιπτώσει. Το ΕΛΚ χαιρετίζει τη συμφωνία της Γενέβης από την Κομισιόν στα πλαίσια του ΠΟΕ για τις εισαγωγές μπανάνας από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Κατόπιν τούτου, να προσθέσω επίσης ότι αντιλαμβανόμεθα τη σημασία της συμφωνίας. Τώρα τελείωσε στα πλαίσια του ΠΟΕ μια μακρά διένεξη που για δέκα ετίες ε, μας ε, δημιουργούσε πρόβλημα γιατί υπήρχαν διακρίσεις σε βάρος των παραγωγών μπανάνας από τη Λατινική Αμερική προς όφελος των χωρών ΑΚΕ. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσουμε πολύ σύντομα αν συμφωνούμε, αν συγκατατιθέμεθα στην ιστορική αυτή συμφωνία. Η γνώμη μου είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δείξει ότι είναι υπεύθυνο παίκτη, ικανός να λαμβάνει καλέ αποφάσεις στο διεθνές εμπόριο και να δώσει πράσινο φως σε αυτή τη συμφωνία. Σύμφωνο επίσης ε, με τον εκπρόσωπο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τον κύριο Αρίφ, που είπε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ακόμα. Και Υπάρχει και μια άλλη πλευρά της υπόθεσης αυτής που είναι ότι θα υπάρξουν και σαφή ιτημένοι και σαφείς ζημίες μετά την απελευθέρωση της αγοράς μπανάνας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μου είναι σαφές ότι μειώνοντας τα ε, ε, δασμολογικά εμπόδια θα πρέπει να φροντίσουμε να μην αφανίσουμε τομείς και κλάδους που κατά παράδοση έπαιξαν τόσο σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ε, ρόλο σε κάποιες περιφέρειες της Ευρώπης. Τελειώνω, τελειώνω. Να φροντίσουμε επίσης ότι παράλληλα με τα μέτρα απελευθέρωσης του εμπορίου θα πρέπει να διασφαλίσουμε τους παραγωγούς μπανάνας για να μπορέσουν να παραμείνουν στην αγορά και να συνεχίσουν τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Κύριος Μάτο, δύο λεπτά. Ένα λεπτό, Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι λυπάμαι που άκουσα αυτό Αυτή είναι μια εξαιρετική συμφωνία. Μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμφωνία για την επιτεύξη της Συρίας, όμως δεν είναι μια καλή συμφωνία για τον τομέα της μπανάνας. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα μέτρα αξιολογήσεις του αντικτύπου και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι από τα 176 ευρώ ανατόνο περνάμε στα 114. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μια καλή συμφωνία για τον τομέα της μπανάνας. Έτσι λοιπόν Πρέπει να ζητήσουμε, αναζητήσουμε αντισταθμίσεις, πρέπει να υπάρχουν αντιστάσεις για τον τομέα της μπανάνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αυξηθεί το κονδύλι. Ευχαριστώ. Two minutes, and I mean it. Δύο λεπτά και το εννοώ. Μην ε, στενοχωριέστε, κύριε Πρόεδρε. Όχι, έχω λόγους. Είχα λόγους για να στενοχωριέμαι. Νομίζω ότι η παραγωγή και οι εργαζόμενοι στον κλάδο της μπανάνας, οι αφρικανικές χώρες, οι χώρες της Καραϊβικής θλίβονται και διαφωνούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νέα Συμφωνία. Οι χώρες αυτές είχαν ενθαρρυνθεί εδώ και πολύ καιρό να αυξήσουν την παραγωγή μπανάνας γιατί αυτό θεωρεί το τομέα κλειδί για την ανάπτυξή τους και τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσής τους και την αύξηση της απασχόλησής τους. Ενώ τώρα ε, σε πολλά επίπεδα η Ευρωπαϊκή Ένωση για δικούς της επιχειρηματικούς σκοπούς τράβηξε το χαλί κάτω από την προσέγγιση αυτή της πολιτικής. Ακολουθεί άλλη πολιτική. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις για πολλούς φτωχούς και μικρούς παραγωγούς σε αυτές τις χώρες. Η νέα συμφωνία αδιαμφισβήτητα είναι υπέρ ε, των πολύ μεγάλων πολυεθνικών εταιριών φρούτων που κυριαρχούν στην παραγωγή στην Κεντρική και Λατινική Αμερική και είναι σαφές ότι οι προτάσεις της Κομισιόν που τώρα τίθενται σε εφαρμογή συνδυάζονται με την πίεση υπέρ μεγαλύτερης απελευθέρωσης του εμπορίου στην Κεντρική και Λατινική Αμερική σε σχέση με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με Κολομβία και Περού και σε σχέση με τους στόχους των ευρωπαϊκών μεγάλων επιχειρήσεων να ε, μπει με μεθόδους εκφοβισμού σε τομείς εμπορίου, υπηρεσιών κλπ. στη Λατινική και Κεντρική Αμερική. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε άλλο δρόμο με βάση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και το σεβασμό στο περιβάλλον. Όλα αυτά τώρα αντιμετωπίζονται πολύ αρνητικά από τη Νέα Συμφωνία. Τέσσερα λεπτά, κύριο Σαρίφ, για τελικά σχόλια. Δεν ναι, ναι, έχω ιδιαίτερε παρατηρήσει. Νομίζω ότι η Φραντσόσκα εξέφραζε τη θέση μα. Το θέμα δεν είναι εδώ τώρα αν επιχειρούμαστε για τη συμφωνία. Η συμφωνία ΠΟΕ προέκυψε κατόπιν συγκρούσεων ιστορικών και αυτό θα, ούτως ή άλλως θα έπρεπε να επιληθεί οι χώρες ε, ΑΚΕ θα συναντήσουν ε, πάρα πολλές δυσκολίες ε, όταν το 72% των εισαγόμενων μπανανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται ήδη από τη Λατινική Αμερική και κυριαρχούσαν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, ιδίως η Τσικίτα. Εδώ θέλουμε να έχουμε πραγματικά αντισταθμιστικά μέτρα και για τις ε, χώρες ΑΚΕ αλλά και για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές ε, και το ότι δεν αντιποκρίνεται η Κομισιόν σήμερα σε αυτά, αυτό με λυπεί. Εδώ ολοκληρώνουμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Θα επανέλθουμε για να εξέταση ε, του σχεδίου της έκθεσης ε, έχει προγραμματιστεί για την 1η και 2 Δεκεμβρίου και θα ξαναρχίσουμε τις συζητήσεις μας στις 3 με μια δημόσια κρόαση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Σας ευχαριστώ και καλή σας όρεξη.